Bien je propose que nous commencions notre réunion. Bonjour à Kalimera sas, sas proteinon archisoume te synedriasis. Al momento que la soñe señora y a la ha terminado. Gracias. Euh je vous propose que nous commencions notre Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του πρέδρου μας που έχει αναγκαστεί να παραμείνει στο κράτος του και που κανονικά θα πρέπει να έρθει το απόγευμα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος. Θα σας ενημερώνω κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να χαιρετήσω τους υπαλλήλους του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους βοηθούς μας, ε, τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και τη γραμματεία μας. Και θα έχετε λάβει τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της 17ης Νοεμβρίου 2011 και Εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το μεσημέρι, μάλλον μέχρι το τέλος της μέρας, ε, θα θεωρηθεί πως εγκρίνονται. Να επιστήσω την προσοχή σας ε, σε διάφορα θέματα. Οι γλώσσες καταρχήν ε, επαρκούν για την πολιτική έκφραση των βουλευτών είμαστε και στο ε, web. Υπάρχει απευθείας μετάδοση στο web. Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε μικρόφωνο να παίρνετε το μικρόφωνο που βρίσκεται στα αριστερά σας. Προτείνω λοιπόν να στραφούμε αμέσως στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην Ουγγαρία, πέντε χρόνια μετά από την προσχώρηση. Την εφαρμογή των, την, μάλλον την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τον έλεγχο και την εποπτεία. Θα δώσω το λόγο στην Ίγκερ Γκρέσλε που είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήμουνα, αν θέλετε, επικεφαλή τη αντιπροσωπεία. ήταν ε, πολύ επιτυχή η επίσκεψη στην Ουγγαρία και όπω πάντα αξίζει τον κόπο να συζητάμε με αντιπροσώπους των κρατών μελών. Διαπιστώσαμε ότι όταν καταφτάσαμε στην ε, Ουγγαρία, η Ουγγαρία βρίσκεται σε μια φάση μεταρρύθμισης σε ό,τι αφορά το δημόσιο κλάδο. Δηλαδή, βλέπουμε καινούργια άτομα των οποίων οι εργασίε είναι πλέον διαφανείς. Είδαμε ότι πρόκειται για μια ε, κυβέρνηση η οποία έχει αλλάξει με την κατάργηση, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά μόνο το δημόσιο κλάδο, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για το τι θα σημαίνει αυτό για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Είπαμε με μεγάλη σαφήνεια λοιπόν ότι δεν μας συναρπάζουν ιδιαίτερα οι μεταρρυθμίσεις και δεν θέλουμε ασφαλώς να μπλεχτούμε στα εσωτερικά ενός κράτους μέλους, αλλά θέλουμε να υπάρχει και μια νομική βεβαιότητα ως προς τους ε, ομολόγους μας. Ιδιαίτερα επειδή το πρόβλημα αυτό το έχουμε θέσει επανειλημμένα. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούν και όλοι οι συνάδελφοι. Είδαμε ότι η Ουγγαρία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της κρίσης, τα οποία όμως και αντιμετωπίζει. Είδαμε επίσης ότι πρόκειται για ένα κράτος μέλος, το οποίο ασφαλώς αφέ αυτό αντιμετωπίζει πολιτικά προβλήματα εσωτερικά σε ό,τι αφορά την πολιτική κατάσταση της χώρας. Νομίζω ότι ήταν επιτυχής η επίσκεψη αυτή, γιατί είδαμε ότι το κράτος μέλος βάλει κάθε προσπάθεια να προωθήσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να κάνει μια επαγγελματική διαχείριση όλων των προγραμμάτων. Ε, ασχοληθήκαμε με θέματα εσωτερικής ε, διοργάνωσης κατανομής των πόρων στα διαφορετικά ταμεία. Εκτενώς ασχοληθήκαμε με το κρατικό ταμείο, το γεωργικό ταμείο και είδαμε ότι η Ουγγαρία, όπως και η πλειοψηφία των κρατών μελών, δεν έχει δεν θέλει να προβεί σε βαθιά αγροτική μεταρρύθμιση. Και να ρωτιόμαστε προ προς τα που οδεύει αυτή η αγροτική μεταρρύθμιση. Είδαμε λοιπόν στα μεγάλα έργα ότι όπου υπήρχαν ατασφαλίες υπήρχε θέληση να παραμεριστούν. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της συνεργασίας τη καταπολέμηση της απάτης σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Όλαφ και είδαμε ότι υπάρχει ε, μια υπηρεσία αντίστοιχη για την επικοινωνία με, τον, με την Όλαφ αλλά δεν είναι πάντα ε, ενήμερη για το τι ε, προτείνει και τι ε, συστήνει η Όλαφ. Αυτό θα ήταν μια πρόταση. Επίσης κατατίσαμε μια σχετική έκθεση να ευχαριστήσω τη γραμματεία για την έκθεση αυτή, η οποία λοιπόν ε, έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις, τις συστάσεις μας. Νομίζω ότι ήταν σωστό το ότι ταξιδέψαμε στην Ουγγαρία και παρά το γεγονός ότι η Ουγγαρία δεν είναι στην κορυφή των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ήταν σίγουρα σωστό να γίνει επίσκεψη στην Ουγγαρία ως ένα νέο κράτος μέλος. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την διοργάνωση του ταξιδίου που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ίγκε, για την έκθεση αυτή. Υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι να προσθέσει? Η Κομισιόν. Merci. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εικόνα που προκύπτει από την ε, κοινοβουλευτική αποστολή ε, στην Ουγγαρία συμπίπτει με την εικόνα που έχουμε εμείς στην Κομισιόν για την διοίκηση της Ουγγαρίας, η χώρα αυτή, για τη χώρα αυτή γενικότερα ε, ο διοικητικός μηχανισμός έχει περάσει από πολλές μεταρρυθμίσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει κάποιους κινδύνους βέβαια, πράγμα που έχουμε εμείς εντοπίσει και έχουμε ενημερώσει πολλές φορές. Ο νέος ε, ε, διοικητικός μηχανισμός ωστόσο φαίνεται να λειτουργεί με ικανοποιητικό τρόπο και να προχωρεί με ικανοποιητικό τρόπο στη διαχείριση των υποθέσεων. Η Ουγγαρία είναι μια χώρα η οποία ε, χαρακτηρίζεται από κεντρική διοίκηση, κεντρική διαχείριση, κεντρικό έλεγχο και εποπτεία των διαρθωτικών ταμείων. Υπάρχει ένας μηχανισμός που συνδέεται άμεσα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και άρα αυτό είναι το κεντρικό σημείο για τη διαχείριση των ε, κονδυλίων των διευθυντικών ταμείων. Αυτό έχει τονιστεί και όταν εντοπίστηκαν προβλήματα, τα προβλήματα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης ε, από πλευράς των Ουγγρικών αρχών και άνευ θα πρέπει να πούμε ότι η Κομισιόν θεωρεί πως η διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί ε, άμεσα δράση στην Ουγγαρία. Και βεβαίως θα πρέπει η εθνική νομοθεσία να προσαρμοστεί με την κοινοτική. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και ως εκ τούτου οι διαδικασίες έχουν ε, βελτιωθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν κάποια προβληματάκια, αλλά πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις ε, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, θα πρέπει να διαπιστώσουμε Υπάρχουν λοιπόν μερικές, ε, μερικά προβληματάκια που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα για τον ανταγωνισμό στις δημόσιες συμβάσεις, στις κρατικές προμήθειες και κάποιες φορές ε, δεν γίνεται απόλυτα επαρκής ε, χρήση των κοινοτικών πόρων, δηλαδή υπάρχει υπερβολικό κόστος για κάποια έργα, για κάποιες επενδύσεις, σπανίως. Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως η Ουγγαρία είναι μια χώρα που απορροφά αποτελεσματικά τα κορδίλια των διευθυντικών ταμείων, δηλαδή τα αποτελέσματά της είναι ανώτερα από τον μέσο όρο, αν συγκριθούν με αυτά των άλλων χωρών που είναι αντικείμενο παρέμβασης των διευθυντικών ταμείων. Είναι μια χώρα που έχει κάνει καινοτόμε δράσεις σε πολλούς τομείς. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω τα όσα έχει κάνει η Ουγγαρία στο θέμα της χρηματοπιστωτικής ε, λογιστικής είναι η χώρα που χρησιμοποιεί ευρύτερα αυτά τα μέσα έχει φτιάξει μια πλήρη δομή που χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να τεθεί σε εφαρμογή και να αρχίσει να λειτουργεί αλλά που σήμερα δείχνει ενδιαφέροντα αποτελέσματα ο αντίκτυπος για τις ε, Ε, στην οικονομία είναι σημαντικός όπως γνωρίζουμε και προφανής ήδη. Είμαστε σε κάποια αρχική φάση βέβαια γιατί αυτά τα μέσα χρειάζονται κάποιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αρχίσουν να αποδίδουν. Πάντως είναι κάτι το θετικό. Κάτι άλλο θετικό είναι η εφαρμογή και διαφόρων ολοκληρωμένων δράσεων που αφορούν είτε το αστικό περιβάλλον είτε το ενίπεθρο ή τους πόλους ανάπτυξης ε, ώστε να υπάρξουν ε, συνεργασίες και επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της στήριξης των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν το πλαίσιο, αυτό, αν και υπάρχουν κάποιες σκιές, γενικά είναι ρόδινο. Η Ουγγαρία κάνει αποτελεσματική χρήση των ιστορικών ταμείων. Αυτή είναι η εκτίμηση της Κομισιόν. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Οράν. Είστε τμηματάρχης της, της Κομισιόν για την Ουγγαρία. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συναδελφό Γκρέσλε για την έκθεση αυτή. Πρόκειται για μια πολύ ξεκάθαρη ε, έκθεση και έχει νόημα να ε, μεταβαίνουμε σε μια χώρα που δεν βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιότητων μας γιατί Εκεί μπορούμε να δούμε το τι συμβαίνει ακριβώς σε περιπτώσεις που δεν αναμένεται η παρουσία μας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά για την απορροφητικότητα, τη δυνατότητα απορρόφησης της Ουγγαρίας. Και τότε τα βασικά προβλήματα, τις βασικές αιτίε πρόκειται για συνήθεις αιτίε. Το συνηθισμένο θέμα του ποιο κάνει τι, πώς ορίζουμε τη συνεργασία μεταξύ κομισιών και κρατών μελών, Όλα αυτά λοιπόν είναι κλασικές περιπτώσεις. Θα ήθελα να σημειώσω θετικά για την Ουγγαρία ότι μπορεί και έχει δείξει διάθεση να μάθει. Και αυτό προκύπτει και από την έκθεση. Αναφέρονται τα όσα έχουν βελτιωθεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν ε, χώρες που κάνουν διαρκώς τα ίδια λάθη και δεν είναι διτεθειμένες να προσαρμοστούν. Στην επόμενη απαλλαγή θα υπάρξει ε, μια νέα κλιμάκωση, γιατί αν τα κράτη-μέλη μας είπε, για παράδειγμα, ο Επίτροπος ε, μετα, ότι η Πολωνία είναι εξαιρετική παράδειγμα για το πώς ε, απορροφούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και η Ουγγαρία τα πηγαίνει επίσης πάρα πολύ καλά. Γιατί λοιπόν η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τα πηγαίνουν καλά. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος και να μην εργαζόμαστε με διακοπές αλλά με αναστολές. Αναστολές των πληρωμών για τις χώρες εκείνες που διαρκώς σφάλουν, όπου ξέρουν ότι δεν πρόκειται να επιτελέσουν το έργο τους όπως, πρόκειται, όπως ε, πρέπει. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Γκρέσλε. Ευχαριστώ κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Γκρέσλε για την έκθεσή της και για τις συστάσεις της. Θα ήθελα μόνο να ρωτήσω δύο, δύο πράγματα σε σχέση με την επίσκεψη. Κυρίως προς την Κομισιόν απευθύνομαι. Και σχετίζονται με τα όσα είπε ο κ. Χατζημαρκάκης που και έχουν ε, ε, σημασία. Το ελεγκτικό συνέδριο μας είπε ότι υπήρχαν προβλήματα με το, την Ουγγαρία. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν συνέβη στην Ουγγαρία. Δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα, αλλά Φυσικά και οι συνάδελφοι μίλησαν για την δυνατότητα απορρόφησης και μία από τις δυνατότητες ήταν ακριβώς αυτή. Τότε αυτό αποτέλεσε και ιδιαίτερο κριτήριο για την Ισπανία. Το θέμα λοιπόν είναι ποια είναι η σχέση μεταξύ της επίσκεψης αυτής και των όσων μας αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο για τη χώρα αυτή. Και κατά δεύτερον, τι γίνεται μετά εργαλεία διαμόρφωσης. Γιατί και εγώ είμαι από αυτούς που προασπίζω, προασπίζω την ε, υποστήριξη των ε, ε, εργαλείων αυτών. Το θέμα λοιπόν είναι σε ποιους τομείς λειτουργούν τα εργαλεία για την χρηματοοικονομική διαμόρφωση. Σε ποιους τομείς λοιπόν λειτουργεί η κατάσταση. Euh, ευχαριστώ. Η κυρία Γιάννα Σένα αναφέρθηκε στο ηλεκτρικό συνέδριο. Πώς το ηλεκτρικό συνέδριο θέλει να σχολιάσει. Όχι. Α, Chris Vaughan. Uh, uh, uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την έκθεσή της, ιδίως τις συστάσεις που αναφέρονται στην έκθεση. Αλλά διαβάζοντα την έκθεση είδα ότι υπήρχαν δύο θέματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Γιατί δεν καλύπτονται από καμία από τι συστάσεις. Το ένα είναι οι δημόσιε προμήθειε και το ερώτημα με είναι εάν οι συνάδελφοι θεωρούν τώρα τα πράγματα είναι εντάξει σε αυτό το τομέα. Και το δεύτερο είναι το θέμα του οργανωμένου εγκλήματο που αναφέρεται στη σελίδα 11 τη έκθεση. και λέγεται για το οργανωμένο έγκλημα ότι μια προβλεπόμενη τροπολογία της, του ποινικού κώδικα της Ουγγαρίας που θα τεθεί σε ισχύ το 2012 και Είναι μια πρόταση που δεν είναι πάρα πολύ σαφής και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η νέα αυτή νομοθεσία θα αντιμετωπίσει την κατάσταση καλύτερη ή χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη της αντιπροσωπείας μας που πήγαν στην ε, Ουγγαρία και μάλιστα παραμονή των διακοπών όπου οι περισσότεροι βουλευτές ε, το μόνο που σκέφτονται ήταν πώς θα φύγουν διακοπές. Ε, ακόμα πιο θερμά συγχαρητήρια λοιπόν. Πιστεύω πως ε, έτσι καταργείται ο μύθος που λέει ότι στις χώρες της νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κοινοτικά κονδύλια ε, υποαπορροφώνται ή, εν περιπτώσει, χρησιμοποιούνται χειρότερα από ό,τι στις χώρες της ε, παλαιάς Ευρώπης. Τέτοιου είδους στερεότυπα δυστυχώς εξακολουθούν να ακούγονται και να ισχύουν ε, αλλά όπως αυτή η αποστολή στην Ουγγαρία συμβάλλει στην κατάργηση αυτών των μύθων. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κανένας άλλος βουλευτής να πάρει το λόγο και θα ήθελα να επανέλθω ως Ευρωβουλευτής. Παρα, παρακαλώ, κυρία μου. Σας ευχαριστώ. Δύο λόγια για να απαντήσω στα ερωτήματα που αφορούν τα απορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου για τον προϋπολογισμό από το Ταμείο Συνοχής και δύο λόγια για τις δημόσιες συμβάσεις. Όσον αφορά την Ουγγαρία, ακούσαμε και από μάλλον και από πλευράς της Κομισιόν με τα πρώτα προγράμματα ΕΣΠΑ το 2002-2003 συμμετείχαμε εκεί και κάναμε έλεγχο και κάτι που προέκυψε ήταν η μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων τότε στο πρώτα προγράμματα ΕΣΠΑ. Κάναμε ελέγχους για αυτές τις δημόσιες συμβάσεις ε, αλλά αυτό που είδαμε θα πρέπει να σας πω ήταν αλλαγή ότι δηλαδή οι Ουγγρικές αρχές ε, δέχτηκαν πρόθυμα τις διορθώσεις που τους προτείναμε από την πλευρά της Κομισιόν και δέχτηκαν να αλλάξουν τους κανόνες και την εφαρμογή αυτών πιο συγκεκριμένα. Πιστεύω πως ένα από τα προγράμματα τα οποία ελέγχθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούλιο, όπως αυτό της ε, ε, επεξεργασίας λιμάτων της Βουδαπέστης ήταν ένα από τα έργα τα οποία έγιναν μετά από την αποδοχή από τις Ουγγρικές Αρχές των Αλλαγών που αναφέραμε και ε, αναφερόταν και στον έλεγχο του 2007 από το από το ελεγκτικό συνέδριο. Όπως σας είπα, εξακολουθούμε να βρίσκουμε προβληματάκια, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει βούληση για αλλαγή σε αυτές τις διαδικασίες. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να προσθέσω κάποια στοιχεία σε σχέση με τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα των ε, μέσων που χρησιμοποιήθηκαν εκεί είναι στοιχεία τα οποία διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης ε, την περασμένη εβδομάδα. Ο αριθμός των εταιριών μέχρι στιγμής που έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτές, δηλαδή που έχουν λάβει επιχορηγήσεις με αυτή την έννοια, τις έχουμε φτάσει σε αυτές, έχουν λάβει κάποια χρηματική βοήθεια, είναι 5.200. Τα ποσά που έχουν ε, εκχωρηθεί για όλα τα μέτρα συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ε, για την κεντρική ε, Ουγγαρία που είναι περιοχή σύγκλησης είναι 232 εκατομμύρια. Και αυτό θα πρέπει να συγκριθεί με το σύνολο του κονδυλίου που είναι 750 περίπου εκατομμύρια. Δηλαδή πάνω από το 25% έχει ήδη απελευθερωθεί και δοθεί, αλλά Περισσότερα ακόμα πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά νομίζω πως εν γέννη είναι ικανοποιητική η κατάσταση, δεδομένου ότι υπάρχει και ένα χρονικό διάστημα που χρειάζεται να περάσει μέχρι ότου να θεσπιστούν αυτού του είδους τα μέτρα. Υπάρχουν ε, μια ολόκληρη σειρά προγράμματα για προϊόντα, για κεφάλαια κινδύνου και ούτω καθεξής και φυσικά μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία σε σχέση με όλα αυτά τα αποτελέσματα. Γυρία Αγιάλα, ναι, θέλω μόνο να ζητήσω κάτι, μια διευκρίνηση από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που μίλησε για το σχέδιο για το πρόγραμμα μάλλον ε, του έργου για την επεξεργασία λιμάτων της Βουδαπέστης. Θα ήθελα να μου πει λοιπόν αν οι Ουγγρικές αρχές δέχτηκαν τις διορθώσεις της Κομισιόν και στην έκθεση στη σελίδα 16 λέει ότι οι Ουγγρικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν αυτά τα ποσά και σε άλλα προγράμματα επιλέξιμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης. Ότι δηλαδή τα περισεβούμενα ποσά μπορούν να δοθούν σε άλλα παρόμοια προγράμματα. Μέχρι ότου ναι. να συνονεθεί η Επιτροπή για να δώσει την απάντηση, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να θέσω μια ερώτηση για να απαντήσει η Κομισιόν. Μιλήσατε για δημόσιες συμβάσεις κύριο Ράνη και για βελτιώσεις, αλλά όλες αυτές οι υποθέσεις έχουν προκύψει και στον τύπο. Και ένα σύνολο ευρωπαϊκών εταιριών έχουν εκφράσει την έκπληξή τους για την λειτουργία, θα έλεγα, της διοίκησης επιτόπου. Βεβαίως, για την χορήγηση των ε, δημοσίων έργων, την ανάθεση μάλλον των δημοσίων έργων, αλλά και όσον αφορά τη μονομερή ε, καταγγελία συμβάσεων. Εκεί η Κομισιόν μπόρεσε να κάνει κάτι. Υπήρξε κάποια διαμεσολάβηση. Πού βρισκόμαστε με αυτές τις συμβάσεις που αφορούν ε, στην ουσία δημόσιες συμβάσεις. Φαντάζομαι πως έχετε όλα τα στοιχεία. Διότι αν θέλετε αυτού του είδους η ε, συμπεριφορά δίνει την εικόνα μιας εσωτερικής αγοράς που δυσλειτουργεί. Άρα λοιπόν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες πλήττονται από τέτοιου είδους συμπεριφορές ε, είναι αρνητικό. Τι έκανε λοιπόν η Κομισιόν για αυτές τις υποθέσεις. Για να μην, για να μην παρεξηγήσετε, όχι για τα ευρωπαϊκά ταμεία που κατάβαλα τι κάνετε, είναι για την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Είναι προφανές ότι υπάρχουν φαιές Ζώνε ε, στη λειτουργία των δημοσίων αγορών στην Ουγγαρία, όπω το είπα και προηγουμένω. Όταν μίλησα για μη αναλογική εφαρμογή των κριτηρίων και διάφορων πρακτικών που οδηγούν στον αποκλεισμό κάποιων επιχειρήσεων. βάση εφαρμογής σε μία αναλογική, όπως είπα, νομοθεσίας. Οι διαδικασίες αυτές δεν μπορούν εύκολα να κατηγορηθούν όσον αφορά την μη νομιμότητά τους. Γιατί υπάρχουν κάποια νομικά κριτήρια που μπορεί κανένας να θεωρήσει ότι έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Εσείς αναφερθήκατε επίσης στα συμβόλαια που καταγγέλλονται κατόπιν. Η Κομισιόν βέβαια δεν έχει αρμοδιότητα οι αρμοδιότητες είναι στα χέρια των διαφόρων υπηρεσιών της λειτουργία τη εσωτερική αγοράς προφανώ. Ε, κοιτάμε βέβαια τι γίνεται με την καλή διαχείριση των διαθετικών ταμείων. Πολλέ φορές ε, χρειάστηκε να παρέμβουμε με ρόλο διαμεσολαβητή αν θέλετε για να διευκολύνουμε τις σχέσεις των δύο ε, μερών Πολλές φορές μπορεί αυτό να θεωρηθεί απόλυτο δικαιολογημένο και πολλές φορές πετύχαμε έτσι μια συμφωνία μεταξύ των συμβαλωμένων μερών η Κομισιόν πραγματικά ανησυχούσε πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη περίοδο που έχω κατά νου. Γιατί η λειτουργία του σχεδίου εξαρτώται από την αβεβαιότητα του κατά πόσον οι συμβάσεις πραγματοποιούνται ως προεβλέπεται ή όχι. Έχουμε λοιπόν μια ένδειξη για την ύπαρξη προβλημάτων και στην περίπτωση αυτή παρακολουθούμε την εξέλιξη και αν δούμε ότι δεν συμβαίνουν τα πράγματα που πρέπει προσπαθούμε να παρέμβουμε. Πρόεδρος, με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά από ό,τι κατάλαβα τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν επλήγησαν γιατί είπατε ότι κάνατε τις διορθώσεις. Η συγκεκριμένη μου ερώτηση ίσως δεν αφορά τη δική σας ε, υπηρεσία, αλλά αυτό που ρωτάω είναι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων της λειτουργίας των εσωτερικών αγορών που φαίνεται ότι έχουν καταπατηθεί και από όσο ξέρω είναι αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να ξεκινήσει τη διαδικασία επιπαραβάση για τις χώρες που δεν εφαρμόζουν σωστά τους ε, κοινοτικούς κανόνες. Γιατί αν τελικά η τοπική συμπεριφορά είναι αντίθετη με τους κανόνες για λειτουργίας αγοράς, πρέπει να δράσει η Κομισιόν. Εγώ θέλω λοιπόν να με διαβεβαιώσετε ότι λειτουργούν οι κανόνες της εσωτερική αγοράς και στην Ουγγαρία. Απάντηση. Φυσικά, μόλις γνωρίσει κάποια παρανομία η Κομισιόν, αντιδρά αμέσως. Αυτό που αναφέρατε εσείς δεν αφορά κάποια παρανομία, στις περιπτώσεις που ξέρω τουλάχιστον, αλλά το θέμα είναι του κατά πόσον οι νόμοι είναι σωστοί. Δηλαδή εφαρμόζονται νόμοι που θα μπορούσε κανένας να θεωρηθούν ως ε, μη αναλογικοί. Δηλαδή οδηγούν σε μια απόφαση που ε, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις αλλά μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη. Είναι ένα πρόβλημα που είδαμε σε ορισμένε περιπτώσει. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να εκτιμήσω το εύρος του προβλήματος. Το σε αυτή την κρίζα ζώνη γιατί δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι παράνομο, αλλά μπορούμε να δούμε κατά πόσον αυτή η νομοθεσία είναι σύμφωνη ή όχι με την ε, σωστή λειτουργία της αγοράς. κυρία Γιάλα Σέντερ, θέλει επίσης μια απάντηση στην ερώτησή σας. Il faudrait renouveler la question. Euh, Μήπως θα πρέπει να επαναλάβετε την ερώτηση. Ναι, πρόεδρε, Σα ευχαριστώ. Αναφερθήκα στην περίπτωση το δάτων τη Βουδαπέστης υπήρχε εκεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχετε ήδη μια λύση γιατί η Κομισιόν είχε κάνει μια πρόταση για κάποια μέτρα. Εγκρίθηκαν από την Ουγγρική κυβέρνηση αλλά φαίνεται ότι τώρα οι πόροι χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση για κάποιες άλλες διαδικασίες ή όχι. Νομίζω ότι είναι συνήθις αυτή η διαδικασία όταν γίνονται δηλαδή διορθώσεις χρησιμοποιούνται οι πόροι αλλού. Είναι σωστό αυτό? Ναι, για το θέμα αυτό πράγματι. Η διόρθωση που πρότεινε η Κομισιόν τότε ήταν 25% ενός πολύ σημαντικού ποσού για τα λίματα του Βουδαπέστης. 250 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Το 25% λοιπόν οφείλεται σε μη σωστή εφαρμογή της διαπραγματευτής σας διαδικασίας. Εάν θυμάμαι σωστά ήταν γύρω στα 40 εκατομμύρια και έχετε δίκιο ότι όταν ο κράτος μέρος αποδεχτεί τη διόρθωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια αυτά που ελευθερώνονται για άλλες ε, επιλέξιμες ε, δαπάνες, για άλλα στοιχεία μέσα στο φάκελο αυτό. Αν δεν δέχονται όμως την διόρθωση, η διόρθωση θα ήταν καθαρή από τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Έχετε δίκιο. Πράγματι, δεν βλέπω κανένας να θέλει να υποβάλει άλλη ερώτηση. Η για να ολοκληρώσει έχει το λόγο. Α, πολύ ωραία αυτή τη συζήτηση, η οποία κατέληξε τώρα πόσα προβλήματα έχει μια χώρα που θεωρείται ότι δεν έχει προβλήματα. Και γι' αυτό ε, συμφωνώ με τον κύριο Χατζηνοκακάκη που είπε ότι δεν ήταν εσφάλμα να πάμε εκεί. Και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να επαγρυπνούμε για κάτι πράγματα. Ε, θα μπορούσε κανένα να καταλήξει και σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αν βλέπει δηλαδή το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εγώ αποφάσισα να το δω μισογεμάτο, αλλά. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Και αυτό που είδαμε συμπεριλάβει και κάποια πράγματα που δεν μπορούσαν να μας εξηγήσουν. Παραδείγματο χάρη για την επεξεργασία των λιμάτων υπάρχουν πάρα πολλές ε, ε, πτυχές χρηματοδότησης αλλά δεν λένε παραδείγματος χάρη τι πρόκειται να γίνει με τις λάσπες του βιολογικού καθορισμού ή παραδείγματος κάνει και το σχέδιο Τζέρεμι και αυτό είναι ένα ανησυχητικό ε, σχέδιο τώρα τι θα γίνει με το Τζέρεμι στην Ουγγαρία πώς θα το εκτιμήσουμε κλπ όλα αυτά είναι πράγματα που μα ενδιαφέρουν Θεωρώ ότι αυτή η μικρή συζήτηση με την Κομισιόν κατέδειξε πόσα πράγματα και η ίδια Κομισιόν δεν γνωρίζει. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικό πρόβλημα. Ότι η υπηρεσία ε, παρουσίαση των, των ε, αποτελεσμάτων στην Κομισιόν από πλευρά των χωρών είναι ένα σημαντικό θέμα που δεν γίνεται πάντα. Και πρέπει να επιμένει η Κομισιόν. Και αν ξέρουμε, μπορούμε να αντιδράσουμε νομίζω, αλλά πρέπει να ξέρουμε. Και στην κοινοβουλευτική επιτύχη έχω να πω κάτι που με προβλημάτισε. Δηλαδή συζητήσαμε με τους εθνικούς βουλευτές τι κάνουμε με τις εκθέσεις του Ουγγρικού Ελεκτικού Συνεδρίου. Και είδαμε ότι δεν υπάρχει καμία κατανομή της εργασίας. Άρα δεν ασχολείται κανένας με τις εκθέσεις αυτές. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα να στραφώ προς τους ε, συναδέλφους που ε, θεωρούν ότι εάν δεν γίνει πλήρης εξέταση είναι καλά. Όχι, εγώ θα σας πω ότι η Ουγγαρία βρίσκεται σε ισχυρότερη μοίρα από ότι εμείς και ίσως πρέπει να σκεφτούμε μεταξύ των συντονιστών εάν θα πρέπει να εισαγάγουμε μία μόνιμη παρουσίαση από τις περιφέρειες, ούτως ώστε να έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας και να ξέρουμε ποιος ασχολείται και ποιος δεν ασχολείται και τι ε, συνέχεια θα πρέπει να δώσουμε. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχαν, όλοι ήταν δεσμευμένοι για το θέμα αυτό, αλλά θα σας αποκλείσω, αλλά μεταξύ των τεσσάρων μελών και του ενός εθνικού βουλευτή είχαμε 7 υπαλλήλους της Κομισιόν. Ε, δεν ξέρω, δηλαδή ξέρουμε ότι παρέχει προσωπικό η Κομισιόν, πρέπει να μας το δείχνει έτσι ξεκάθαρα κάθε φορά. Για να στηρίξω αυτή την ιδέα της κυρίας Γκρέσλε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μονάδα στο κοινοβούλιο που να ασχολείται με τα εθνικά κοινοβούλια. Και εάν συμφωνήσουν οι συνονιστές θα μπορούσαμε να έχουμε στο μέλλον μια πλήρη συνεδρίαση για κάποια θέματα με τους εκπροσώπους αυτούς των εθνικών κοινοβουλίων. Θα μπορεί να γίνει αυτό σε επίπεδο επιτροπών ή παραδείγματο χάρη για να ακολουθήσουμε αυτά που είπε και η κυρία Γκρέσλε. Πρόεδρο, μου φαίνεται ότι η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αν θέλουμε τα εθνικά ελεκτικά συνεδρία να περάσουν στην αλυσίδα του ελέγχου, θα μπορεί η επίδραση αυτή στα κρατημένη να γίνει μέσω των εθνικών βουλευτών. Και γι' αυτό, όσον αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, τον έχουμε εμεί στην εργασία Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, είναι πάρα πολύ καλή. Και ευχαριστώ την κυρία Γιάννα Σέντερ που υποστήριξε αυτή την πρόταση. Λοιπόν, μπορούμε νομίζω τώρα να κλείσουμε αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο περίπου 4. Αλλά πριν περάσουμε στο σημείο 4, θα ήθελα να χαιρετήσω μία αντιπροσωπεία από το Massif Central της Γαλλίας που ήρθε να ακούσει με πάθος τις εργαστές της Επιτροπής ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου. Είναι από τη δική μου εκλογική ε, περιφέρεια. Μπορούμε να τους χειροκροτήσουμε κιόλας. Συνήθως ε, το κάνουμε αυτό στην Ολομέλεια της ε, επιτροπές, δεν ε, χειροκροτούμε, αλλά καλό ήταν. Τώρα περνάμε τέλος πάντων στο σημείο παραθμών 4. Ειδική έκταση ελεκτικού συνεδρίου, η αποδεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα συνδρομή Ευρωπαϊκή Ένωση που διοχετεύεται μέσω οργανώσεων των ΗΕ σε χώρε που πλήττονται από συγκρούσει. Έχουμε μια έκθεση εξαιρετικής ποιότητας που θα μας παρουσιαστεί από το ηλεκτρικό συνέδριο, ο κύριος Κάρελ Πίνγκστεν. Euh, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ακρόαση σας ενώπιον της Επιτροπής μας και του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, γιατί σας επρότεινε το δικό σας ε, κράτος να είσαστε στην επόμενη θητεία μέλος του Ελεκτρικού συνεδρίου και τύχατε της θετικής ψήφου και θέλω να σας χαρώ γι' αυτό. Je ne pas de... Δεν προδικάζω βέβαια του αποτελέσματος της Ολομέλειας και του Συμβουλίου των Υπουργών, αλλά θέλω προς το παρόν να σας συγχαρώ και να σας δώσω το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Και σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Τι να σας πω, α? τι περιμένετε να σας πω. Οπωσδήποτε θα ήθελα να ευχαριστήσω. Monsieur le député de cette commission pour la confiance τα μέλη της Επιτροπής σας για την εμπιστοσύνη που εξέφρασε προς το άτομό μου. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι έκανα λάθος. Έκανα λάθος γιατί όταν είδα να έρχεται όλη αυτή η αντιπροσωπεία, εμείς θεωρούσαμε ότι είναι από τα Ηνωμένα Έθνη οι κύριοι και οι κυρίες αυτές, αλλά είναι παραπάνω, ανώτεροι, από τη δική σας εκλογική περιφέρεια εκπρόσωποι. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να τους χαιρετήσω εδώ παρέμβαση του Πρόεδρου εκτός μικροφώνου, δυστυχώς. vous Ξέρετε ότι εξετάζουμε σήμερα τη δεύτερη έκθεση για τα Ηνωμένα Έθνη. Στην αρχή το ηλεκτρικό συνέδριο είχε προβλέψει μία μόνο έκθεση και την χωρίσαμε ε, στα δύο για να κερδίσουμε χρόνο. Αυτή η έκθεση γιατί έγινε, για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος, τα ποσά προβλέπονται και που αυξήθηκαν σημαντικότητα. Το 2001 υπήρχαν 144 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεση του ΟΗΕ. Το 2009 935 όμως εκατομμύρια. Πάρα πολύ σημαντικά ποσά λοιπόν και σημαντικότητας αυξήσεις. Δεύτερον, ο τρόπος διαχείρισης με τον οποίο υπάρχουν ε, ε, προβλήματα πολλές φορές, δηλαδή η κοινή διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διεθνείς οργανώσεις. Τρίτη αιτία συγκεκριμένο ενδιαφέρον που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως αυτή εδώ η Επιτροπή για, την, για τον έλεγχο αυτό πριν εξετάσω τα τρία θέματα που θα μας απασχολήσουν, έχω να πω ότι πρόφατο και η λεκτέα μας και εμείς ξέρουμε ότι όταν χρησιμο... διατίθενται τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου στα Ηνωμένα Έθνη για να τα δαπανίσουν σε περιοχές σύγκρουσης τα χρήματα αυτά δαπανούνται κάτω από πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, εν τελευταία αναλύση η, Κομισ... το... η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και οι δαπάνες αυτές γίνονται κάτω από πολύ δύσκολες και εξαιρετικές συνθήκες. Τέσσερα σημεία θέλω να θέξω κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο είναι το πεδίο ελέγχου. Δεύτερον, η ενημέρωση, η έλλειψη ενημέρωσης. Θα είμαι σύντομο. Τρίτο, θα ήθελα να αναφέρω δύο παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά, αλλά δύο θα ήθελα να αναφέρω και κατόπιν θα ήθελα να ολοκληρώσω με κάποια μηνύματα. Θα ήθελα First point, Ξεκινήσαμε Ξεκινήσω με το πρώτο θέμα, λοιπόν, το πεδίο εφαρμογής, ε, το πεδίο που κάλυψε ο έλεγχος. Τρεις χώρες κάλυψε λοιπόν ο έλεγχος, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Σουδάν. Δεκαεννέα project, δεκαεννέα έργα, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στο προσάρτημα, το παράρτημα των ε, εγγράφων. Τι εκτιμήσαμε λοιπόν, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, και τη βιωσιμότητα των έργων. Των οκτώ έργων μάλιστα που έχουν ολοκληρωθεί, που έχουν υλοποιηθεί. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τα 19 έργα αυτά αντιπροσωπεύουν το 80% και πλέον των ευρωπαϊκών πόρων που δαπανήθηκαν μέσω των Ηνωμένων Εθνών στις τρεις χώρες αυτές. Άρα δεν πρόκειται για ένα τυχαίο δείγμα, όχι, αντιπροσωπεύουν 80% και πλέον των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν στην περίοδο 2006-2008. Να πω επίσης ότι στην αρχή ελπίζαμε ότι θα μπορούσαμε να διεξάγουμε ελέγχους επιτόπου σε κάθε μία από τις τρεις χώρες, αλλά τελικά επισκεφτήκαμε μόνον το Σουδάν Μετέβη μάλιστα εγώ ο ίδιος εκεί για λόγους ασφαλείας ήταν αδύνατον να μεταβούν ομάδες στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Αυτά σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, το πεδίο που κάλυψε ο έλεγχος. Δεύτερο στοιχείο τώρα, η έλλειψη πληροφόρησης. Το ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα αυτό, κατά την ε, ακρόασή μου. Σε πολλές περιπτώσεις δεν ήμασταν σε θέση να λάβουμε επαρκείς σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες. Άρα, τελικά, οι ελεγκτές μας δεν συνέλεξαν όλα τα τεκμήρια που μπορούσαν και που ήθελαν να συλλέξουν. Αυτό ασφαλώς επηρέασε την αξιολόγηση και την εκτίμηση και στις τρεις κατηγορίες, και για την αποτελεσματικότητα και για την αποτελεσματικότητα και για τη βιωσιμότητα. αλλά όπως αναφέρεται στην έκθεση ήταν πολύ προβληματική η κατάσταση σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα, όπως αναφέρεται την παράγραφο 44, γιατί σε 7 από τα 9 project τελικά δεν μπόρεσε να ελεγχθεί η αποδοτικότητα. Άρα θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει α, εκτενείς και αξιόπιστες πληροφορίες από τον ΟΗΕ για να μπορεί να αξιολογεί τα έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Και αυτό δεν συμβαίνει για από πολλά από τα έργα. Αυτά ως προς το δεύτερο σημείο. Για το τρίτο σημείο τώρα. Δύο παραδείγματα να σας δώσω που μιλούν από μόνο τους. Θα βρείτε και άλλα πολλά παραδείγματα στην έκθεση και μιλάμε για παραδείγματα πολύ συγκεκριμένα. Θα ήθελα να φερθώ πρόεδρε, στην σελίδα 70, στο πρώτο πεδίο, σε ό,τι αφορά το τμήμα που έχει την επικεφαλίδα άνεπαρκές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τον Νότιο Σουδάν. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό πριν από την ανεξαρτησία. 65% των δαπανών στην τελική έκθεση αναφέρεται ως πρώτερα έξοδα. Πρώτερα έξοδα. Πρώτερες δαπάνες, χωρίς καμία ή αδίποτε άλλη πληροφορία για τη φύση των δαπανών. Μόνο πρώτερες δαπάνες, πρώτερα έξοδα. Φανταστείτε το δηλαδή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς έπρεπε να αρκεστούμε σε αυτές τις πληροφορίες. Αυτό καταδεικνύει πόσο ανεπαρκείς είναι οι πληροφορίες που χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο παράδειγμα, 21 σελίδα, προγράμματα τα οποία δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους. Εκαθάριση Ναρκοπαιδείων στο Αφγανιστάν. Πολύ σημαντικό έργο. Ποια ήταν τα αποσκοπούμενα αποτελέσματα της εκαθάρισης. 26,6 τραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτός ήταν ο στόχος, ο αρχικός για την εκαθάριση. Και τελικά πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα εκαθαρίστηκαν, όχι 26,6, 1,6 μόνο. Άρα νομίζω ότι αντικειμενικά ο στόχος δεν επιτεύχθη. Αυτό καταδεικνύει πόσο ε, περιορισμένη είναι η αποδοτικότητα. Τέταρτο και τελευταίο σημείο τώρα, Πρόεδρε. Κάποια μηνύματα, αν θέλετε να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Γκρέσλε για το εξαιρετικό έγγραφο εργασίας που κατήρτισε. Δεν θα επαναλάβω τα όσα αναφέρει στην έκθεσή της, ούτε θα μπω σε λεπτομέρειες για τα πολλαπλά απορίσματα, τα οποία όλα α, τα αναφέρει η κυρία Γκρέσλε. Κάποια μηνύματα μόνο θα ήθελα να να Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει καταρχάς να διασφαλίσει ότι υπάρχουν σαφείς στόχοι, επιτεύξιμοι στόχοι για κάθε έργο, οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθούνται και αν κατά πόσο είναι δυνατόν να μπορούν να μετρούνται, να μπορούν να ποσοτικοποιούνται για όλα τα έργα και αυτό μάλιστα προτού δεσμευτούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεύτερο μήνυμα θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα αποδοτικότητας των έργων και στην αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Γιατί δεν αρκεί να διαπιστώσουμε ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες. Αυτό είναι προϋπόθεση. Φυσικά θα πρέπει να είναι επιλέξιμες, αλλά αυτό δεν τα λέει όλα. Τρίτο μήνυμα. Η έκθεση, ε, η πρόοδου, η έκθεση follow-up που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον ΙΕ, θα πρέπει να παρακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εντοπίζονται ενδεχόμενε πηγές προβλημάτων. Και τελευταίο μήνυμα είναι ότι χρειάζονται κατάλληλα μέτρα όχι μόνο για την αντιμετώπιση αλλά και για τον τερματισμό του συνεχικούς προβλήματος της ε, ελπής κατάρτισης εκθέσεων και υποβολής αναφορών από πλευρά του ΟΗΕ. Φυσικά, αναφέρθηκε και πριν από δύο εβδομάδες νομίζω στην Επιτροπή, καλωσορίζω τις πρόσφατες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ιστορικές ε, εκθέσεις ελέγχου και άλλε τέτοιε ενδείξει για μεγαλύτερη διαφάνεια από πλευρά του ΟΗΕ. Αλλά θεωρούμε ότι στη φάση αυτή που ελέγχουμε τα νέα αυτά έγγραφα, τα νέα τεκμήρια, θα πρέπει να διαπιστώσουμε κατά πόσο αρκούν αυτές οι νέες προθέσεις. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Η συγκεκριά μας είναι η Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ. Στην ειδική... Πρόκειται για τη δεύτερη ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου τα τελευταία χρόνια για την ε, κοινή αρρωγή μέσω διεθνών οργανισμών. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι και τον Φεβρουάριο του 2009 υπήρξε και έγινε μια αποστολή ε, στην ΟΗΕ, στην οποία και συμμετείχα για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Τώρα, ακούγοντα ότι κοιτάμε δύο, τρεις δύσκολες χώρες, ε, Σουδάν, Αφγανιστάν και νομίζουμε ότι και Ιράκ. Το έγγραφο εργασία αυτό το έθεσα στο ε, επίκεντρο, αν θέλετε, των προσπαθειών μας να λάβουμε πιο πολλές πληροφορίες από τον ΟΗΕ. Να θίξω τα γενικά προβλήματα συνεργασίας με τον ΟΗΕ, με τον Παγκοσμία παγκόσμιους οργανισμούς γενικά τα βασικά προβλήματα της συνεργασίας αυτής τα έβαλα στο επίκεντρο της έκθεση γιατί φυσικά αναγνωρίζω ότι έχουμε ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτές τις τρεις χώρες αλλά διαπιστώνουμε ότι γενικά χρειάζεται καλύτερη ευθύνη, καλύτερη, καλύτερες εξηγήσεις από τον ΟΗΕ. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, πολλές ε, υποσχέσεις έχουμε ακούσει, αλλά τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Ωστόσο, η πίεση αποδίδει καρπούς. Ο ΟΗΕ πρόσφατα εξασφάλισε πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιστορική έκθεση ελέγχου σε ό,τι αφορά έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίεσης την οποία ασκήσαμε στις συστάσεις μου τώρα. Θα ήθελα να τονίσω κάποια ζητήματα τα οποία εύκολα μπορούν να επιτευχθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως πριν από το λογιστικό έτος θα μπορούσε να μας πει πόσα χρήματα σκοπεύει να διαθέσει στον ΟΗΕ. Αυτό ε, έχει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι επιτρέπει και στον ΟΗΕ και στις άλλους οργανισμούς ε, να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, γιατί πολλές φορές μου έχουν αναφέρει οι οργανισμοί αυτοί ότι ε, αυτοί ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας τους δυσκολεύει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κονδύλια ευρωπαϊκά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα, καλύτερο σχεδιασμό, καλύτερο προγραμματισμό και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Αλλά η ευελιξία δεν μπορεί να ισχύει παντού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση μια ολόκληρη χώρα. Ένα πρόβλημα ιδιαίτερο είναι τα καταπιστευματική μία πολλών χορηγών. 60% των ε, δαπανών περνάνε μέσα από καταπιστευματικά ταμεία πολλών χορηγών. Στα τρία από τα 19 αυτά έργα της, ε, που εξετάσει το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν ξέρουμε δηλαδή αρκετά στοιχεία για τα μεγάλα αυτά έργα, για το μεγάλο αυτό όγκο των ταπανών. Είχα στη διάθεσή μου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια ε, εσωτερική έκθεση της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα τέτοιο ταμείο και τα αποτελέσματα τα συμπεριέλαβα και στις συστάσεις μου. Το Εθνικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι μέσω των έμεσων ε, εξόδων, μάλλον ότι για τα έμεσα έξοδα, για τα διοικητικά έξοδα, δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες. Και έτσι τα διοικητικά έξοδα αυτά εγκρίνονται χωρίς έλεγχο. Μήπω το λεκτικό συνέδριο θα μπορούσε να καταρτήσει ένα ειδικό, μια ειδική έκθεση σε ό,τι αφορά τα καταπιστευματικά ταμεία αυτά, γιατί μιλάμε για μεγάλα ποσά. Οι συνάδελφοι που ήταν στην ε, περιοχή που επλήχθη από το σεισμό θα θυμούνται ότι μας είπαν ότι αυτό το ταμείο διέθετε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά τελικά ορατά ήταν μόνο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Άρα θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να καταρτήσει ελεγκτικό συνέδριο ε, μια ειδική έκθεση για τα ταμεία αυτά. Νομίζουμε ότι πολλά θα διαπιστώσουμε. Να επενθυμίσω επίσης ότι αυτό παίζει και ρόλο σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική τάξη. Τα παλιά θέματα, πρόσβαση ε, για το ελεγκτικό συνέδριο, πρόσβαση γενικά σε έγγραφα Αυτά πάντα έπαιζαν ρόλο και εξακολουθούν να παίζουν ρόλο και το λέω αυτό με κάποια απογοήτευση ότι προχωρούμε με ρυθμούς χελώνας στα θέματα αυτά. Γι' αυτό να παρακαλέσω το ελεγκτικό συνέδριο να αποτυπωθούν αυτές οι δυσκολίες και στην έκθεση απαλλαγής. Οι συστάσεις μου περιλαμβάνουν πάντα και τις παλαιότερες συστάσεις το θέμα είναι αν δεν υπάρχει βελτίωση θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι είναι καλή η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, είναι σκόπιμη, αλλά στην όλη ιστορία, σε ό,τι αφορά τα παλαιά προβλήματα, πρέπει να σα πω ότι δεν μου αφήνει πολύ καλή εντύπωση το γεγονό ότι δεν σημειώνεται πρόοδο στα παλιά αυτά θέματα. Να σα ευχαριστήσω γιατί ήταν πολύ εκτενή οι συζήτησή μου με το ελεγκτικό συνέδριο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα Ηνωμένα Έθνη ασφαλώ και με κάποιους οργανισμούς των ΗΠΑ συγκεκριμένα, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι περιμένουμε ε, πιο πολλέ εξηγήσει από το απλά να μα λένε πόσο περίπλοκο είναι ο κόσμο. Σα ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στου εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων, η Κομισιόν, ο κύριο Σμίτ, ίσω έχει να μα πει δύο λόγια. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν καλωσορίζει την έκθεση και θα περιορίσω τις παρατηρήσεις μου σε κάποια σημεία τα οποία θίγει και η συγκίτρια στις συστάσεις της και τα 10 σημεία στις σελίδες 6 και 7 της έκθεσής της. Καταρχήν στο σημείο 4 η βασίζει το θέμα της καταγραφής και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κοκομπού για τη στήριξή της σε αυτό το θέμα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε συμφωνήσει με το Ηνωμένα Έθνη τον Απρίλιο πέρσι ένα νέο ε, μια νέα έκθεση μάλλον μάλλον ε, κατευθύνες γραμμές για το τι θα πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις εκθέσεις ε, οπωσδήποτε γιατί βασιζόμαστε σε αυτές. Και υπάρχει ένα θέμα ποιότητος και ε, κυρότητος. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι θα εφαρμόζουμε αυτές τις κατευθύντες γραμμές για ένα χρόνο και μετά θα επανέλθουμε στην άνοιξη του 2012 για να δούμε αν αυτές οι νέες κατευθύντες γραμμές είχαν τα τεχνικά αποτελέσματα και θα αναφέρουμε στο Κοινοβούλιο τα πορίσματά μας. Δεύτερο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι η αποτελεσματικότητα που αναφέρεται και στο θέμα ε, του εισηγητή, στην έκθεση του εισηγητή ε, στο σημείο 26. Είναι αλήθεια πως η, Κομισι... η της Κομισιόν βασικά είναι εκ των προτέρων και αφορούν τους πυλώνες, να δούμε δηλαδή κατά πόσο πληρούνται οι ε, κανόνες για να ξεκινήσουμε και είναι κάπως δύσκολο σε τέτοιες χώρες να παρακολουθήσουμε μετά τον αντίκτυπο. Είναι προφανές όταν μιλάμε για χώρες όπου η Κομισιόν δεν έχει καν αντιπροσωπεία. Αυτό συνέβαινε στο Νότιο Σουδάν μέχρι πρόσφατα. Θα ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία στη Τζούμπα. Ε, στις άλλες δύο χώρε ήταν πολύ δύσκολη πρόσβαση επί Φυσικά και έχουμε αυξημένες προσδοκίες και έχουμε κάνει μια πρόταση στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό 57,5 που εισάγει αυτή τη δήλωση αξιοπιστίας για την κοινή διαχείριση. Ελπίζουμε πως αυτό θα υιοθετηθεί και έτσι θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το θέμα της αξιοπιστίας από τους εταίρους που εφαρμόζουν τα προγράμματα. Να μιλήσω και για το θέμα των ημερών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο. Γιατί σε 7 η συγκίτρια μιλά για ρεαλιστικά χρονικά πλαίσια. Αυτό είναι θέμα που δεν αφορά μόνο τα όσα κάνουμε με το ΝΟΙΕ, αλλά όλες τις περιπτώσεις όπου εργαζόμαστε υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες και θα υπήρχε ίσως βάση για να παρατείνουμε την δράση μας, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες και αν θέλουμε να επιτύχουμε τους αρχικούς στόχους και να, έτσι να προστατεύσουμε την επένδυση, καλύτερο είναι να παρατείνουμε λίγο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δράση, το έργο και να μην χάσουμε την επένδυση. Και αντιστρόφως ανάλογα μπορεί να υπάρχουν καλοί λόγοι για να το σταματήσουμε. Και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στα προγράμματα συνεργασίας με τον ΟΗΕ. Θα έχουμε δείκτες κλειδιά για την απόδοση, όπου θα παρακολουθούμε τις διάφορες μας, με τις διάφορες μας αντιπροσωπείες για να δούμε αν υπάρχουν συνήθιστες καθυστερήσεις σε κάποιες περιοχές. Να ολοκληρώσω με ένα θετικό μήνυμα σε σχέση με την πρόσβαση στον έλεγχο και πάλι πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το εκτελεστικό διευθυντήριο της UNICEF, UFCD και ούτω καθεξής που έχουν συμφωνήσει να αποκαλύψουν τις, εσωτερικούς, τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου. Ε, είναι ένα θετικό μήνυμα αυτό θετικό το κλίμα συνεργασίας μας με τον ΟΗΕ και φυσικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκμεταλλευτούμε τα όσα μπορούμε να μάθουμε από αυτές τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου του ΟΗΕ. Αυτά και φυσικά θα απαντήσω σε ερωτήσεις αν υπάρξουν μετά. Ε, ευχαριστώ, Κύριε Κυρία Γέλα, έχετε έτσι το λόγο. Και Σα presidente. Sí, yo también eh, felicitar, desde luego, a la colega Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε για την έκθεσή της. Ε, ε, ε, αυτή είναι η ζωή μας. Μέσα στη χρηματοδότηση. Οι διεθνείς οργανώσεις δεν έχουμε μόνο το Ηνωμένα Έθνη. Στο σημείο 2.2 το λέει και η κυρία Γκρέσλε στην εκθεσή τη, όπω το είπε και ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν καλή πρόοδο, νομίζω, επιτελέσει. <clears throat> και το χαιρετίζουμε αυτό ιδιαίτερα. Θα ήθελα τώρα, στραφόμενοι προς την Κομισιόν, να ρωτήσω ποιο είναι το χρονοδιάκαμα που προβλέπετε. Οι, οι εσωτερικές αυτές εκθέσεις της Κομισιόν σε ποια χρονική κλίμακα δίνονται, γιατί δεν ξέρω επίσης αν υπάρχουν και όλες τις υπηρεσίες, Ορισμένε μου λείπουν. Πού πρέπει λοιπόν να ασχίσουμε πίεση για να συμμετάσχουν όλες οι υπηρεσίες και ποια είναι τα παραδείγματα που μπορούμε να έχουμε. Δεύτερο, επίσης τρεφόμουν προς την Κομισιόν. Και προς το ηλεκτρικό συνέδριο βέβαια. Οι προτάσεις που υπάρχουν στην έκθεση είναι ελιστικές γιατί με όλη αυτή τη συζήτηση για το ποσοστό σφάλματος και τους κινδύνους που ενέχονται είχαμε κατά και αυτά τα σχέδια τα οποία προωθούνται βάσει πολιτικών αποφάσεων σε περιοχές ε, για τις οποίες συμφωνούν βέβαια οι πολίτες της Ένωσης να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά υπάρχουν από εκεί και πέρα τα προβλήματα του ελέγχου. Δηλαδή εξ είναι πολύ δύσκολο, ε, εξ post ε, εκ των υστέρων δηλαδή είναι επίσης προβληματικός ο έλεγχος. Λοιπόν, αναρωτιέμαι κατά πόσον αυτές οι προτάσεις είναι ρεαλιστικές. Γιατί τα ποσοστά σφάλματος είναι σημαντικά και θα ήθελε έπρεπε ίσως να τα δούμε και μέσα στα πλαίσια των δηλώσεων ex όχι εξάτε και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται συνεχώς τουλάχιστον εγώ το είδα δύο-τρεις φορές ε, στην έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Ιράκ δύσκολη κατάσταση δεν είμαστε αντίθετοι με την βοήθεια αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν συμπληρωματικά προβλήματα και δεν ξέρω κατά πόσο η Κομισιόν έχει κάτι να μας πει, γιατί αναφέρεται εκεί ότι το 70% των δαπανών ήταν περιτές. Και είναι δύσκολο η Κομισιόν τώρα να αιτιολογήσει τους πόρους αυτούς ή και να τους επανεισπράξει. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Και κάτι άλλο. Στρεφόμενοι προς τον κύριο Πίνσεν. είδα ότι έδωσε κάποιε πληροφορίε στη συνάδελφο Γκρέσλε σήμερα το πρωί. Θα ήταν καλό πληροφορίε αυτέ να δοθούν σε όλου του συναδέλφου. γιατί πιστεύω ότι αυτέ οι διμερείς ε, ε, πληροφορίε είναι κάποιε προβληματικέ. Ευχαριστώ κύριο Χατζημαρκάκη. Εγώ αντίστροφα θα ήθελα να εγκομιάσω τον κύριο Πίξεν για την έκθεσή του. Σπάνια ακούμε τόσο σαφή, ανοιχτή και καλά δομημένη έκθεση σε μια προφορική παρουσίαση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την τόσο επιτυχία αυτή παρουσίαση σας. Παρ' αυτά έχω και προς τον ίδιο αλλά και προς την Κομισιόν μία ερώτηση αρχής. Εξετάζοντας ότι οι πόροι ε, δίνονται με τρεις ε, μεθόδους ε, το διεθνούς οργανώσεις. Δηλαδή καταρχήν σε συγκεκριμένη σχέδια. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να είναι και απολύτως ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση στις περιπτώσεις αυτές. Δεύτερον, δίνονται σε κάποια ταμεία των δωρητών και τρίτον στο γενικό προπολογισμό των ε, οργανώσεων του ΟΗΕ. Αυτό αναφέρεται εδώ στην εκθεσή σας. Λοιπόν, αναρωτιέμαι αυτό κατά πόσο να αποφέρει και το ρωτώ αυτό γιατί ε, βλέπουμε από διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λιγότερα χρήματα. Τα κράτη-μέλη είναι έμεσα μέλη του ΕΕ. Δεν ξέρω, σας ρωτώ αυτό, είναι θέμα αρχής. Μήπως θα πρέπει να δίνουμε χρήματα για συγκεκριμένα σχέδια που να αναφέρεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μέσω του προϋπολογισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον οποίο κατά βάση είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη. Και ήθελα να πω να περιοριστούμε σε αυτά που είμαστε ορατοί και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν από μόνα τους να, να δράσουν μέσα του τα κρατημέλη που είναι μέσα, ε, μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Ευχαριστώ κύριος Γκανιέρ. Ja, die Frage, wollen Το κατά πόσο θέλουμε τα χρήματα αυτά να διανύμονται μέσω των ε, υπηρεσιών του ΟΗΕ είναι σημαντικό θέμα και θα πρέπει να εκτιμήσουμε ακριβώς τα μειονεκτήματα και τα πλέον Και προσπάθησα να το δω αυτό πρώτον το Ηνωμένα Έθνη μπορούν να πάνε εκεί που δεν μπορεί να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η σημαντική διαφορά. Στα πλαίσια της δικής μου έκθεσης αναρωτήθηκα κατά πόσο θα έπρεπε να πάω στο Αφγανιστάν. Όταν μου είπανε στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, αλλά εμεί δεν βγαίνουμε από το συγκρότημα αυτό στην Καμπούλ γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Ε, και είπα τι να κάνω. Ε, ποιος ο λόγος δηλαδή να κινούμε με τεθωρακισμένο αυτοκίνητο από τεθωρακισμένο ε, ξενοδοχείο στο ε, τεθωρακισμένο αν θέλετε συγκρότημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην δω τίποτα επιτόπου πραγματικά ή τι να πάω. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε επιτόπου τόπου έλεγχους ε, όπως το κάνουν οι Αμερικάνοι που πάνε ας πούμε σε ένα σχολείο, πάνε στο, σε ένα σχολείο μια μονάδα των Marines, ε, μετράει τους υπολογιστές, ξαναφεύγουν με το ελικόπτερο, αλλά δεν ξέρουν οι υπολογιστές αυτές την επομένη εξακολουθούν να παραμένουν και που τους μετρήσανε. Κατά γενικό κανόνα μπορούμε να πάνε εκείνοι εκεί που τα πάμε εμείς. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα περικόψουμε τα κονδύλια μας στο Ευρωπαϊκό, στην, ε, στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά αυτό θα περιορίσει όμως την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, ε, το θέμα της ορατότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχω διαφορετική άποψη ε, από την εξώτιμη κυρία εισηγήτρια. Εάν δίνουμε τα χρήματά μας σε ένα διεθνές ταμείο, το κάνουμε για διάφορους λόγους. Ή τα δίνουμε μέσω του ΟΜΙΕ για τους λόγους που σας είπαμε ότι μπορούν να μπουν σε το μίσο που δεν μπορούν να πάνε. Και δεύτερον, ότι έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ε, επίδρασης. Το κατά πόσον είμαστε αιρετοί ή δεν είμαστε, είναι δύσκολο να πάω σε ένα σχολείο και ε, να πάω στο σχολείο και να σας πω εντάξει αυτό το σχολείο χρηματοδοτήθηκε από ένα διεθνές ε, ταμείο αλλά να μου πείτε ποια είναι τα κεραμίδια που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όχι. Το, μόνο που μπορούμε να πούμε ήταν ότι τα χρήματά μας ήταν το 100% των πόρων και ότι οι πόροι αυτοί πήγαν εκεί και μπορούμε να δούμε πραγματικά πόσο είναι η δική μας συμβολή. αλλά δεν μπορώ να πω ότι θέλω να δω ακριβώς ποια είναι η σύμβολη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο, οι ανεπαρκές πληροφορίες. Προσπάθησα να το κατανοήσω παρόλο που είμαι μόλις από το 2009. Εγώ κατάλαβα ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε πολλά προβλήματα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μέλος του ΟΗΕ είναι υπέρ. Δεν ξέρω αν τα κράτη-μέλη θα ήταν υπέρ. Και θα ε, κατέληπαν ορισμένα από τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Αλλά βέβαια το ο τώρα δεν μπορεί να μας ε, αντιμετωπίσει σαν ένα πλήρες μέλος. Έχω κατανόηση γι' αυτό βέβαια. Το πρόβλημα είναι πως θα έχουμε επαρκείς πληροφορίες. Και έχω σχετικά και ένα ερώτημα προς τον, ε, το ηλεκτρικό συνέδριο και προς την Κομισιόν. Εγώ από ό,τι κατάλαβα Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο οργανώσεων όσον αφορά το τι γίνεται με τα, φα, φα, τα έγγραφα αυτά του ΟΗΕ. Τι γίνεται δηλαδή με τη συμφωνία με τον ΟΗΕ. Η Κομισιόν λέει όλα καλά. Το ηλεκτρικό συνέδριο λέει δεν αρκούν όμως. Γιατί βάσει των ΦΑΦΑ δεν έχουμε τις επαρκές πληροφορίες. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα άλλαζαν τα πράγματα αν ήταν μέλος ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν, χρονοδιαγράμματα. Οι μη κυβερνικοί μας μα είπαν πολλέ φορέ ότι είναι πολύ σύντομα τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία θα πρέπει να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται, τι διατάξει είναι αυτέ. Είναι πολιτικέ ε, προδιαγραφέ των ε, δωρητών που θέλουν να έχουν γλυκό αποτέλεσμα αλλά δεν είναι ρεαλιστικά. Είναι θέμα της πραγματικής κατάστασης επιτόπου. Από πού προέρχονται αυτές οι προθεσμίες. Γιατί εάν δεν μπορούμε στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές να έχουμε ρεαλιστικές ε, προδιαγραφέ χρονικές πού μπορεί κανένας να βασιστεί σε μια χώρα που βρίσκεται εν μέσω εμφυλίου πολέμου και που δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή. Αυτές οι ερωτήσεις μου και οι ευχαριστίες μου και πρέπει να το πω εκ μιας αρχής ευχαριστίες στον κύριο Πίξτεν του Ελεκτικού Συνέδρου και στην εισηγήτρια. Το η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών γιατί δεν είναι κράτος. Πολύ απλό. Ο κύριος Παλτσίτης, ευχαριστώ πρόεδρε. Διάβασα τα έγγραφα και ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας. Όλα τα κονδύλια τα οποία διαθέτουμε είναι στην αποκλειστική μας ευθύνη ως προς την διανομή τους. Και είμαστε υπόλογοι στα κράτη-μέλη, στις επικράτειές μας, που καλούνται να πληρώσουν το μεριδιό τους στο γενικό προϋπολογισμό. Μία ερώτηση, το σύστημα που ίσχυε παλαιότερα βελτιώθηκε σημαντικά, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει όλη έννοια της απόδοσης ευθυνών και της λογοδοσίας σε ό,τι αφορά τα κονδύλια αυτά. Κινούμαστε αργά. Αναφερθήκατε ελεγκτικό συνέδριο στο άρθρο 57 που αναφέρεται στην πιο αποτελεσματική κοινή διαχείριση. Με την κοινή διαχείριση θα ε, αναλαμβάνετε από τον κάθε φορέα η πλήρης ευθύνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη διανομή των πόρων αυτών. Θα καταρτιστεί ένα καινούριο σύστημα που θα διασφαλίσει την καλύτερη και πιο αποτελεσματική διάθεση των κοντιλίων αυτών. Ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρος, ο κύριο Έρνχάουστον. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε αυτά που είπε ο κύριος Γκάιρ στο πρώτο τμήμα της εισήγησής του και να κάνω μια ερώτηση στο ελεγκτικό συνέδριο. Βρέθηκα στο νότιο Σουδάν και διαπίστωσα ότι είναι εξαιρετική η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Είναι προφανές ότι τα έξοδα και οι δαπάνες στις χώρες αυτές ασφαλώς παρουσιάζουν ελλείψεις, πιο πολλές από τις άλλες περιοχές. Ε, ερωτώ λοιπόν, επί της αρχής ίσως τα ελαττώματα, οι ελλείψεις που διαπιστώνει το ελεγκτικό συνέδριο έχουν την πηγή τους στην μέθοδο κοινή διαχείρισης. Να το θέσω αλλιώς. Η άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τέτοιες περιφέρειες είναι πιο οικονομική και πιο αποτελεσματική. Αυτό ως ερώτηση προς το Ελληνικό Συνέδριο. Euh, donc, est Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη συζήτηση, το ηλεκτρικό συνέδριο θέλει να πει δύο λόγια ίσως. Και η Κομισιόν φυσικά. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais tout d'abord Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας για τον πολύ ενεργό τρόπο με τον οποίο συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. εχω πεντε σελίδε σημειώσει εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάθε ένα από τα σημεία που αναφέρθηκαν. Καταρχήν προς την κυρία Γκρέσελ. Δεύτερον, θα ήθελα να την ευχαριστήσω για το τόσο θετικό της αυτό σχόλιο αναφέρθηκε σε trust funds πολλαπλών δωρητών στο έμεσο κόστος και στο κατά πόσον το συνέδριο θα μπορούσε να κάνει μια ειδική ακρόαση για τα λεγόμενα multi-donor trust funds αυτά. Σημειώθηκε το αίτημα Το κοίταξα και στην έκθεσή Θα το δούμε λοιπόν στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας για το επόμενο έτος. γιατί έχουμε ήδη ακροάσεις που προε... Ε, ελέγχουν συγγνώμη, που προετοιμάζονται και δεν είναι ε, πάντα προφανές το να κάνουμε ένα ειδικό έλεγχο μέσα στα πλαίσια του προγραμματισμού μας. Σημειώνω λοιπόν το αίτημά της Και επί ευκαιρία θα ήθελα να πω στην κυρία Γιάλα ότι έδωσα στην εισηγήτριά σα κάποιε συμπληρωματικές πληροφορίε. Ο στόχο δεν ήταν οι πληροφορίε αυτές να δοθούν μόνο σε εκείνη, αλλά θα μπορούσε να τι διαθέσει ελεύθερα. Φυσικά. Νομίζω ότι αν υπάρχει εισηγητή, είναι ε, φυσιολογικό καταρχήν ο εκπρόσωπος του ηλεκτρικού συνέδρου να στραφεί προς τον ή την εισηγήτρια. Και αυτό αφορούσε την παράγραφο 9 της εκθεσής της. Ήθελα να σας δώσω κάποιες λεπτομερωτικές εξηγήσεις. Δεν ήθελα λοιπόν να σας στερήσω ή οσδήποτε ε, εκμετάλλευση στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν θα σχολιάσω την Κομισιόν. Η Κομισιόν θα απαντήσει από μόνη της. Το άλλο σημείο εκτός από το ενημερωτικό της κυρίας Αγιάλα, κατά πόσον οι προτάσεις αυτές είναι ρεαλιστικές. Και μετά το ύψος του κινδύνου σφάλματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αν έχει κανένας ένα έλεγχο για την ε, χρήση των χρημάτων, εξετάζει την αποτελεσματικότητα την σωστή χρήση και την αηφορία. Αυτό κάναμε. Και εγώ ανέφερα εισαγωγικά στην εισαγωγή μου ότι η Κομισιόν είναι αναγκασμένη να συνεργάζεται με τον ΙΕ κάτω από πάρα πολύ δύσκολες προϋποθέσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι ευθύνη του συνεδρίου να εξετάσει τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου. Είναι ενδιαφέρον το σημείο αυτό συζήτηση μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Καλή συζήτηση ίσως, πάρα πολύ καλή συζήτηση. Ε, όταν γίνει όμως αυτή η συζήτηση, ακόμα και για τις τρεις αναφορές εδώ της έκθεσης, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Πολύ λεπτή η συζήτηση λοιπόν αυτή. Πολύ σημαντικό το θέμα. πράγματα που ίσως δείχνουν πάρα πολύ λογικά για την Κομισιόν, πολύ λογικά για κάποια μέλη του Κοινοβουλίου, ίσως δεν είναι πολύ λογικά για τον ε, φορολογούμενο. Λεπτή λοιπόν αυτή η συζήτηση. Αλλά δεν είναι η συζήτηση που θα γίνει στο ελεκτικό συνέδριο, περσέ. Εμείς σημειώνουμε τις απόψεις του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Εν κατακλείδη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήδη συζητιέται. Για τις παρατηρήσεις του κυρίου Χατζηπαλκάκη, αυτές μάλλον στρέφονται προς την Κομισιόν βέβαια, ο ρόλος των κρατών μελών, δικαίωση και Κομισιόν στον νέο χρηματοδοτικό ε, κανονισμό θα είναι ευθύνη όχι μόνο της Κομισιόν αλλά η Κομισιόν θέλει να διευρύνει τις ευθύνες της και στους άλλους εταίρους. Το θέμα της ορατότητας παραμένει επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Είναι έτοιμο τη συζήτηση αυτό. Θέλετε να έχετε έντονη οραματικότητα, μικρή οραματικότητα. Είναι θέμα αυτό συζήτηση. Και τίνω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι ευρωβουλευτέ θέλουν να είναι μάλλον ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Γκάιερ. Τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να πάνε εκεί που δεν μπορεί να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό αυτό. Και στην κοινή διαχείριση είναι σαφές ότι είναι παρόν σε ορισμένες χώρες στις οποίες δεν είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στην έκθεσή μας δεν λέμε ότι είμαστε αντίθετοι στο να συνεργαστούμε με τον ΟΗΕ. Επουδενή. Αν θέλει να συνεργαστεί με την Ηνωμένα Έθνη ή Κομισιόν, πολύ ωραία. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει αντίτιμα στα χρήματα που καταβάλουμε. θα ήταν πολύ καλό εάν οι πληροφορίε τη Κομισιόν δίνονται εκ των προτέρων. Όπως ανέφερε και η κυρία Γκρέσλι, αν δεν κάνω λάθο. Το πρόβλημα της πληροφορίας που παίρνουμε από το Ηνωμένα Έθνη εξακολουθεί να είναι θέμα συζήτησης και όταν εξετάστηκε η, η δική σα έκθεση πριν από μερικέ μέρες, άκουσα τι παρατηρήσει του εκπροσώπου της Κομισιόν, που έχει το τόσο δύσκολο όνομα, είπε ότι όλα έχουν επιληθεί. Και το ξαναπήγα στο ηλεκτρικό συνέδριο και μίλησα με τον διευθυντή μου, μου είπε όχι, καθόλου. Οι απόψει λοιπόν είναι διαφορετικές και έχουμε ένα καθεστώ παρατηρητή όπου συζητάμε τα θέματα με την Κομισιόν και ο, ο διευθυντή μας ο Φίλιπ Φαντού είναι πάντα παρόν στις ε, συνεντήσεις της ΦΑΦΑ. Θα πρέπει να επιθυμίσω ότι δεν πέρασε πολύ καιρό όταν υπήρχε μία ερώτηση από τους ελεκτές να επανεξατεστεί ο κώδικας επικύρωσης. Λοιπόν, εάν οι ανεξάρτητοι ελεγχθές των Ηνωμένων Εθνών ζητούν επανεξέταση και μάλιστα και διαγραφή της ρήτρα ε, ε σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ ευτυχής με όλες τις πληροφορίες που δίνουν στην Κομισιόν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ. Το θέμα της ΦΑΦΑ λοιπόν παραμένει ανοιχτό και προσυζήτηση. The next um, speaker talked about accountability. Επόμενος ομιλητής ε, μίλησε για την υπολογιστικότητα για το σημείο 7 Αν κοιτάξετε τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό θα δείτε στο άρθρο 1.7.8 ότι υπάρχει αλλαγή του συστήματος που αναθέτουν περισσότερη ευθύνη σε εκείνες οργανώσεις από, που συνεργάζονται με την Κομισιόν και με τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά, εν τελευταία αναλύση, κάποιος θα πρέπει να είναι υπόλογος για μας για τις δαπάνες είναι η Κομισιόν. Ακόμα και αν οι προϋποθέσεις είναι δύσκολες, ακόμα και αν η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί με ε, διεθνείς οργανώσεις. Ε, τελευταία αναλύση εκείνη είναι υπόλογη. Δεν το κρίνω. Αλλά νομίζω ότι όταν δαπανούνται χρήματα του φορολογούμενου θα πρέπει να είναι δυνατό να υπάρχει κάποιος υπεύθυνο. Συγκεκριμένος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό μου φαίνεται. Κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνο. Ο τελευταίος ομιλητής, ο κ. Νάουζη. Είπα βέβαια κάποιες ερωτήσεις επίσης. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με άμεση διαχείριση. Δεν θέλω να ξεπεράσω βέβαια τις ευθύνες μου σαν ένα από τα μέλη του ηλεκτρικού συνεδρίου, αλλά αυτό νομίζω που γκρίνατε ε, ε, στην πλαίσια τη του κ. Γκάιερ πριν από δύο εβδομάδες ήταν πάρα πολύ σοφό. Αφήνεται ανοιχτέ όλες τις δυνατότητες και σε περισσότερες ε, περιπτώσεις όπου υπάρχει παράδειγμα το άρθρο 53 που είναι το σωστό μέσο, άλλε φορέ η έμεση ε, διαχείριση, άλλες φορές ε, ε, από κοινού διαχείριση. Παραμένουν λοιπόν ανοιχτές όλες οι δυνατότητες ανάλογα με τις προϋποθέσεις. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι η καλύτερη λύση που μπορεί να υιοθετηθεί. Λοιπόν, με ρωτάτε κατά πόσο είναι κακό να εργάζεται κανένα μόνο με άμεση διαχείριση ή δεν νομίζω. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πολλών ε, μορφών διαχείρισης. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις και όλα τα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Θα ήθελα εδώ σε αυτή τη συζήτηση να τονίσω επίσης το θέμα της απάτης. Μέσα σε όλους αυτούς τους ελέγχους πιστεύετε είτε στους ελέγχους, ε, οι ελεγκτές της Επικομισιόν, είτε του ελεγκτικού συνεδρίου ότι υπάρχουν απάτες και πώς τις αντιμετωπίζετε αν υπάρχουν. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Um, very briefly, um... Πολύ σύντομα. Να πω στην κυρία Γιάλα Σέντερ ότι το χρονικό πλαίσιο για να λάβουμε τους εσωτερικούς ελέγχους να σας περιγράψω σύντομα ποια είναι η διαδικασία. Τα τμήματα της Επιτροπής κάνουν ε, δείγματα για όλο το είδος, όλα τα είδη ελέγχου, είτε είναι προγράμματα του ΟΗΕ. Σε αυτό το δείγμα έχουμε την ε, διαδικασία της αποστολής επαλήθευσης. Τώρα αυτό που έχουμε με το ΟΗΕ είναι ότι όταν τους ενημερώνουμε ότι θα θέλαμε να επαληθεύσουμε ένα από τα προγράμματα που εκείνοι χειρίζονται, Έχουμε τη δυνατότητα, αντί να κάνουμε επαλήθευση, παίρνουμε την έκθεση εσωτερικού ελέγχου του αν υπάρχει τέτοια, που την έχουν ήδη κάνει εκείνοι δηλαδή. Οπότε βάζουμε σε πράξη την αρχή της ενιαίας, του ενιαίου ελέγχου έχοντας έτσι πρόσβαση στους εσωτερικούς ελέγχους στον Αυτό σημαίνει ότι δεν αποφεύγουμε την επαλήθευση, αντίθετα το χρησιμοποιούμε ως τρόπο του να παίρνουμε τους ε, ελέγχους. Και αυτό στην πράξη λειτουργεί υπηρεσία προς υπηρεσία. Υπάρχει μάλιστα και μια εφαρμογή ηλεκτρονική που μας επιτρέπει με έναν κωδικό να έχουμε πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων. Στην, ε, για τα βασικά προγράμματα χρησιμοποιούμε τον ΟΗΕ όταν ε, Υπάρχει καλύτερη, υπάρχουν καλύτερες δυνατότητες, με της ορατότητας και έχουμε ελέγξει την ε, κατάσταση σε όλες τις συνεδριάσεις της ΦΑΦΑ. Και πρέπει να σας πω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Η επόμενη επιλογή για, που αναφέρατε για τα ταμεία πολυμερών δοτών, δωρητών μάλλον, όταν λάβουμε αυτές τις πληροφορίες, βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση. Ας πάρουμε την περίπτωση του Σουδάν, όπου εκεί κατασκευάζουμε στην ουσία την κυριαρχία μιας τελείως νέας χώρας, δηλαδή απογραφή, ε, καθάριση ναρκοπαιδίων, στήριξη του δικαστικού τομέα. Αυτά όλα είναι πολύτιμα γιατί όλοι οι δωρητές μαζί ε, στηρίζουν όλα αυτά υπό την ομπρέλα, την γίδα του ΟΗΕ την ουδετερότητα του ΟΙΑ, γιατί δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ ευαίσθητο πολιτικά και είναι σαφή ο κίνδυνο να θεωρηθεί πω η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει τη μεριά μια χώρα και όχι της αλληνής. Ε, η χρήση δηλαδή τέτοιων τραστ ε, είναι πολύ θετική σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, τρίτη περίπτωση ε, γίνεται μόνο σε, μία, ε, σε ένα σχέδιο και το γραφείο του ΙΠΑ, εκπροσώπου του ΟΗΕ για τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί δεν δίνουμε καμία άλλη συνεισφορά σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, γιατί όπως είπαμε δεν είμαστε μέλος του ΟΗΕ σχεδόν γίναμε, έχουμε σχεδόν δικαιώματα μέλους στη Γενική Συνέλευση και θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό, αλλά όποτε εγώ δέχομαι ανώτατους διευθυντές του ΟΗΕ, ζητώντας συμβολές τους, η απάντησή τους είναι ότι, ότι ε, θα το εξετάσουμε αυτό όταν θα είστε μέλη του εκτελεστικού σώματος, του Συμβουλίου δηλαδή. Μια διπλωματική, ένα διπλωματικό όχι. Ο κύριος ε, ήταν, ε, ήταν παρόν στην συνεδρίαση ΦΑΦΑ που συμπροέδρευσε μαζί με τον ΟΗΕ. Ζητήσατε ποια ήταν η διάθεση και αν προχωρώνταν τα πράγματα. Ναι, εκεί εξετάσαμε και αξιολογήσαμε το θέμα της ορατότητας θετικά. Συμφωνήσαμε για την πρόσβαση στους ελέγχους. Συμφωνήσαμε για τις κοινέ κατευθυντήριες γραμμές για τις αναφορές. Θα έλεγα λοιπόν πως βοηθάει και πως προχωρά στη σωστή κατεύθυνση η ΦΑΦΑ στον κύριο Ιαν Χάουζερ για το τι θα κάνουμε αν δεν χρησιμοποιούσαμε τον ΟΗΕ σε μια τέτοια περίπτωση όπως το Σουδάν. Τώρα έχουμε αντιπροσωπεία εκεί και έχουμε μια νέα ανεξάρτητη χώρα. Έχουμε λοιπόν την κυριαρχία ενός κράτους που τώρα παγιώνεται. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να στηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις ενός κράτους, ένα κάποιο δικαιωτικό μηχανισμό, οπότε πιθανότητα θα, δοθούν, θα δοθεί στήριξη στο Νότιο Σουδάν και μέσω του ΕΑΛ. Αυτή η επιλογή δεν υπήρχε προηγούμενα, γι' αυτό και τώρα αλλάζει η κατάσταση της βοήθειας, καθώς και η κατάσταση εκεί επί τόπου, αλλάζει. Για τον κύριο Ντί, για την απάτη για τις υποθέσεις που συζητάμε, που λείπτονται δηλαδή, που ελέγχονται από το συνέδριο, κατά, από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν, δεν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις απάτης. Σας, αυτά και σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα, σύντομα. Υπάρχουν τραπεζικές εγγυήσεις όμως οι οποίες ήταν παραποιημένες. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτό να σταλεί στον, στην Όλαφ. Αυτό έλεγε η κυρία Γκρέσλε. Τώρα, για να, τον κύριο Πίνγκστεν, πάντοτε όσον αφορά αυτό το θέμα του κινδύνου, οι πολίτες που πληρώνουν τους φόρους τους, οι οποίοι διαδηλώνουν, είναι αλήθεια ότι δεν θέλουμε να πάμε στο Σουδάν στο Ιράκ, αλλά τέτοιες υποθέσεις είναι που οδηγούν στο ότι ο πολίτης πολύ συχνά άμεσα εμπλέκεται. Όταν δηλαδή θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε, όταν υπάρχουν προβλήματα, παιδιά, γυναίκες κινδυνεύουν ή καταστάσεις ε, σοβαρών ανθρωπιστικών κρίσεων, εκεί πραγματικά μπορούμε να συζητήσουμε για το ποσοστό του κινδύνου ή για τα σφάλματα που έχουν γίνει. Και γι' αυτό δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω. Όταν μιλάμε με τους πολίτες μας, συνομιλούμε με τους συμπολίτες μας, μου λένε ότι δεν υπάρχει πραγματικό ευρωπαϊκό όργανο ελεγκτικό. Μα δεν είναι το ίδιο να παρακολουθεί κανείς ένα πρόγραμμα στη Βουδαπέστη, στη Μαδρίτη, στη Βιέννη και το ίδιο με τα προγράμματα εξουδετέρωσης ναρκών, ναρκοπεδίων στο Αφγανιστάν. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι στη σελίδα 21 και διαβάζω στα γαλλικά πέρα από το μείωση της παιδικής θνησιμότητας για τις οποίες οι διαθέσιμες πληροφορίες φαίνεται να δείχνουν ότι κτλ. Αυτός ο στόχος δηλαδή της μείωσης ε, κατά το ίμιση της θνησιμότητας των παιδιών φαίνεται να είναι το ίμιση αυτού του οικοδομήματος. Οι πολίτες λοιπόν με τους οποίους συνομιλώ καθημερινά μου λένε ότι είναι πολύ διαφορετικός ο στόχος από αυτό που παρουσιάζεται εδώ. Εσείς λέγεται ότι είναι ένα μέσο δημοσιονομικού ελέγχου. Αλλά ο πολίτης σκέφτεται πως δεν το ίδιο. όπως ένα στόχος για το Υπουργείο Οικονομίας ή Οικονομικών στο Σουδάν. Δηλαδή τα ελεγκτικά μέσα θα έπρεπε να μπορέσουν να θέσουν όρια διακρίσεις για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας τι ακριβώς κάνουμε. Ο κύριος Μπαλσίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να έχει απαντήσει στην ερώτηση που είχα κάνει. Ήταν πολύ σαφή η ερώτηση. Είπα ότι έχει αλλάξει η κατάσταση και βλέπουμε ότι η έλεγχη πλέον είναι ανεπαρκείς. Βλέπουμε δε πολλές περιπτώσεις ε, κακοδιαχείρισης και κατάχρησης των κοντιλίων. Ίσως να πρέπει να αλλάξει λοιπόν το σύστημα εκπάτρων και το σύστημα ε, με απόδοσης ευθυνών. Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Ρεκτικού Συνεδρίου γιατί αυτός απάντησε στην ερώτησή μου και είπε ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας νέος κοινός οργανισμός για να απευθύνουμε όλα μας τα ερωτήματα σε αυτόν τον κοινό οργανισμό. Και αυτό σε ό,τι αφορά και την λογοδοσία, σε ό,τι αφορά θέματα του που δαπανήθηκαν τα χρήματα, γιατί πρέπει να τα γνωρίζουμε τα στοιχεία αυτά. Το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης είχε αναβληθεί. Έχουμε λοιπόν λίγο <clears throat> χρόνο. Έχουμε μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων. Σας ξαναδώσω το λόγο, αλλά με συγχωρείτε, αλλά θα επιμείνω για τις απάτες, γιατί είναι θέμα όπου ναι μεν οι συμπολίτε μας δέχονται τα ασφάλματα, αλλά δεν ανέχονται τις απάτες. Να σας πω ότι ναι μεν στο δείγμα της, ε, του συνεδρίου δεν υπήρχε απάτη, μάλιστα, τόσο το καλύτερο, αλλά στις συμβάσεις που, κάνει, που συνάπτει η Κομισιόν και στο, στο, στη Συμφωνία Πλαίσιο Διοικητικής και Οικονομικής Συνεργασίας και το πλαίσιο που προβλέπει, που διέπει τη, τα κονδύλια που χορηγούνται, υπάρχουν ε, λέξεις, υπάρχουν μάλλον ε, καλύπτονται οι αναθέσεις έργων, οι συνεργασίες κτλ. Αλλά δεν υπάρχει λέξη απάτη. Ο εντοπισμός απατών είναι μέσα στο πλαίσιο των ελέγχων ώστε να προληφθεί τουλάχιστον η απάτη. Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο να προληφθούν οι απάτε σε διεθνέ επίπεδο. Όλοι αυτοί οι ελεγχτέ όμω του σα ενημερώνουν εάν διαπιστώσουν απάτη. Υποχρεούνται από την νομοθεσία να σα ενημερώσουν ή όχι. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Μπαλσίτη. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή του για το κατά πόσο υπάρχει με κάποιο σημείο κάποιο βήμα όπου η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και ο ΙΕ συγκεντρώνονται ώστε ο ΙΕ να λογοδοτήσει, θα έλεγα ναι. Αυτό είναι το Συμβούλιο ελεγκτών του ΟΗΕ που συμμετέχουν εκπρόσωποι των διαφόρων κρατών μελών και λαμβάνουν τις εσωτερικές εκθέσεις ελέγχου των υπηρεσιών του ΟΗΕ και αντιδρούν από αυτές τις βάσεις και πάλι επαναρχόμαστε στο ότι η Κομισιόν δεν είναι μέλος του ΟΗΕ επισήμως και άρα δεν συμμετέχει σε αυτό το ελεγκτικό συμβούλιο αλλά όπως αναφέρθηκε ε, ήδη τώρα έχουμε πρόσβαση στις ίδιες αυτές εκθέσεις και έτσι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ότι ε, είμαστε μέρος αυτού του ελεγκτικού μηχανισμού. Ζητώ συγγνώμη αν και πάλι δεν, δεν απαντώ στο ερώτημά σας. Ε, ε, τώρα, κύριε Οντή, φυσικά ο ΙΕ υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις όπως όλοι μας οι εταίροι να μας αναφέρουν περιπτώσεις απάτης και οι ίδιες διαδικασίες για την ανάκτηση ε, των κονδυλίων ισχύουν. Οι απάτες, λοιπόν, μάλλον τα κονδύλια μπορούν να ανακτηθούν από κάποια υπηρεσία του ΙΕ όπως και από οποιοδήποτε άλλο εταίρο μας. κυρία να σας πω ότι τα ταμεία πολλαπλών χορηγών βασίζονται στο δεδομένο, στο γεγονός ότι δεν έχουμε τεκμήρια και κοιτώντα τα, τα έγγραφα στον πίνακα. Ähm, Abbildung Nummer Στην εικόνα 6 και στην εικόνα 4 σε 40% των κονδυλίων δεν έχουμε τεκμήρια. Αυτό είναι το ουσιώδες ε, στα ταμεία πολλαπλών χορηγών. Και θα ήθελα να πω, το θέμα δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά των ταμείων αυτών, το θέμα είναι πώς γίνεται η διαχείριση των ταμείων αυτών και πώς θέλουμε να γίνεται η, να γίνεται η διαχείριση. Δεν θέλω να μου δείξουν ε, ποιο κεραμίδι είναι το δικό μου, ποιο κεραμίδι έχτισα εγώ, αλλά θέλουμε να ξέρουμε τι ποσοστό χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε έργο. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερες απαντήσεις και θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η συζήτηση, γιατί όταν με ρωτάτε το value for money, τι να σας πω δεν έχω ιδέα. Αυτά για τη διεθνή συνεργασία και αγαπητοί συνάδελφοι κατά πόσον, μάλλον όσο ε, ρωτάμε από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού κατά πόσον δαπανήθηκαν μόνο οι πόροι και όχι γιατί δεν απανήθηκαν, νομίζω δεν θα πετύχουμε τίποτα παραπάνω. Μου κάνει εντύπωση η συζήτηση. Είναι σωστή και βοηθάει και ίσως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βγάλει τα χαρτιά της και να τα δείξει πάνω στο τραπέζι. Να μας πει ότι, για παράδειγμα, να παραδεχτεί ότι ξέρει πολύ λίγα για την κατάσταση επιτόπου, γιατί δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι, γιατί η κατάσταση ασφάλειας είναι δύσκολη. Να ξέρουμε ότι δίνουμε αυτά τα χρήματα με μια ελπίδα μόνο να πιάσουν τόπο. Στην φάση αυτή όλα είναι δυνατά. Στο Αφγανιστάν ε, γράφουν οι εφημερίδες στην Αμερική ότι βγαίνουν τα χρήματα αυτά και διοχετεύονται εκτός Αφγανιστάν τελικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν φυσικά οι κίνδυνοι, αλλά ασφαλώς και πρέπει κάτι να κάνουμε στις χώρες αυτές, αλλά να σταματήσουμε να έχουμε ψευδεστήσεις, γιατί υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλές περιπτώσεις ε, απάτης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει και δεν βρήκαμε ούτε μία περίπτωση απάτης να διώξουμε, αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί το πρόβλημα είναι ότι οι κανόνες είναι έτσι φτιαγμένη που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φροντίζει για τίποτα γιατί δεν γνωρίζει τίποτα. Θα πρέπει να αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τη δαπάνη των κονδυλίων αυτών για να ξέρει πώς δαπανούνται. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν πολύ λίγοι συγκεκριμένοι κανόνες για τις διαδικασίες αυτές. Merci, euh, Σας ευχαριστούμε. Με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνουμε την εξέταση του σημείου 4. Α, κύριε Γκάγερ, συγγνώμη. Σα ευχαριστώ για τι διευκρινήσεις, Ινγε. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό συμφωνούμε. Φυσικά όλοι. Τι θέλουμε. Οι οργανισμοί είναι οι οργανισμοί αυτοί, όπω η Παγκόσμια Τράπεζα, να αναλάβουν ένα συγκεκριμένο ρόλο και τις ευθύνε του, να μας πούν πού δαπανούνται τα χρήματα και γιατί δαπανούνται τα χρήματα. Δεν θέμα μάλλον το κατά πόσον μπορούμε να δούμε τι ποσοστό δαπανήθηκε από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την πραγματοποίηση ενός έργου είναι ένα άλλο θέμα η συζήτηση αυτή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση λογοδοσίας. Κάτι άλλο, κατά πόσον συμφωνούμε με τον εσωτερικό έλεγχο του ΟΗΕ και της, και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα αποδεχόμαστε τα στοιχεία αυτά όπως τους δικούς μας ελέγχους ή θέλουμε και δικά μας, δικό μας έλεγχο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το ότι δεν ξέρουμε τίποτα, δεν συμφωνώ. Έχουμε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεγάλους καταλόγους για έργα στα οποία έχουν δαπανωθεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Από την έκθεση για το Αφγανιστάν, αν μπορώ να, να πω ότι υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει ένα θετικό στοιχείο είναι ότι αυτά τα χρήματα που βγήκαν τελικά εκτός Αφγανιστάν δεν ήταν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Γιατί δεν δώσαμε άμεσες ε, βοήθειες. Δεν υπήρχαν δηλαδή άμεσα κονδύλια, ενώ οι Αμερικανοί τα παρουσίασαν πράγματα ότι πλήρωσαν πολύ ακριβά αυτή την αφελή τους προσέγγιση για τις, άμε, για τις άμεσες βοήθειες τα οποία τα χρήματα χάθηκαν στη συνέχεια μετά την ε, Δηλαδή τι, θα δώσουμε 5 ευρώ στον αγρότη και θα το πούμε «Σε παρακαλώ όμως, μην καλλιεργήσεις άλλη ηρωίνη». Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει δώσει προσοχή στη σωστή διαχείριση και στη σωστή δαπάνη των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν είναι όλα τέλεια. Αλλά το ότι δεν ξέρουμε που έχουν πάει τα χρήματα, εγώ το αμφισβητώ. Για το Αφγανιστάν τουλάχιστον μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ε, τρεις ε, ε, έρευνες της Όλαφ σε εξέλιξη στην παρούσα φάση. Η μία έχει να κάνει με μια ΜΚΟ με, μια αυγανική υπηρεσία η οποία προσλάμβανε μόνο μέλη της οικογένειας, της Η κατάσταση θεωρώ ότι εκεί είναι πιο θετική και νομίζω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στα σημεία που μπορεί να υπάρξει βελτίωση και εκεί να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Ζητά το λόγο το ελεγκτικό συνέδριο. Θέλετε τώρα. Να διευκρινίσω μόνο ότι είπα ότι δεν έχουμε καμία ιδέα για το value for money. Το θέμα της αποδοτικότητας των ε, κονδυλίων, κοιτώντας ε, τα στοιχεία που μας χορηγεί το ελεκτικό συνέδριο, μόνο σε αυτό το συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στο ελεκτικό συνέδριο. Ναι, Πρόεδρε. Ε, είχαν ακόμα ερωτήσεις σε δύο βουλευτές και θα ήθελα σύντομα να απαντήσω. Αν μπορώ να, απαντήσω, να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση. Κοινή, κοινός θεσμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο oh yeah. Είναι μια δυνατότητα, κύριε Μπαλασίτη, αλλά τότε η Κομισιόν πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και αν η Κομισιόν αναλάβει μια οποιαδήποτε πρωτοβουλία, εμεί θα την εξετάσουμε και θα δώσουμε το σχόλιο μα. Αλλά δεν είναι δική μας ε, υπόθεση η, πρωτοβουλία, η ανάληψη πρωτοβουλία. Κυρία Γιάλα Σέντερ, κίνδυνο, ποσοστό κινδύνου και ποσοστό ασφάλματο. Πολύ σημαντική συζήτηση και ευαίσθητη, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου δεν μπορούμε να πούμε Ιδού τι είναι αποδεκτό ως ποσοστό κινδύνου ή ποσοστό σφάλματος και σε αυτή την περίπτωση είναι θέμα της Κομισιόν να αναλάβει πρωτοβουλία, να το συζητήσει με το Κοινοβούλιο και να φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά σας καταλαβαίνω πολύ καλά ότι όταν δαπανώνται χρήματα στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, ε, στο Νότιο Σουδάν, δεν είναι σαν να δαπανούμε χρήματα εδώ σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Έχετε απόλυτο δίκιο αλλά είναι ένα θέμα που πάλι δεν αφορά το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο. Αντίθετα, όταν αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 21, εδώ πιστεύω ότι πρέπει να το διαβάσετε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, τι λέμε εδώ, όταν μιλάμε για value for money, μιλάμε για τρία πράγματα. Και το τελευταίο εδώ είναι αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα. Αν δεν έχουμε δηλαδή αποτελέσματα. Τι λέμε στο παράδειγμα. Αν θέλετε ε, ε, των υστέρων να επαληθεύσετε αν έχετε αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο κίνησης, ε, baseline. Αν πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να μοιράσουμε στα δύο, να μειώσουμε κατά το ίμιση το ποσοστό θνησιμότητας, μα τότε θα πρέπει να έχουμε καταρχήν την βάση, ποιο είναι το αρχικό επίπεδο, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να κρίνουμε αν επιτεύχθη ο στόχος ή όχι. για την παιδική θνησιμότητα και ήταν ξεκάθαρο η Κομισιόν πρότεινε ένα συγκεκριμένο στόχο να τον μειώσει κατά το ίμιση, αυτό ήταν σαφές αλλά για άλλα σημεία δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν υπήρχαν κάποια αριθμητικά στοιχεία και αυτό που ζητάμε από την Κομισιόν είναι να λέει ξεκάθαρο στο Κοινοβούλιο ορίστε, θέτουμε κονδύλια στη διάθεση του ΟΗΕ στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Νότιο Σιδάν, οπουδήποτε. Και το σημείο εκκίνηση είναι αυτό και το αποτέλεσμα στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε είναι φυσικά καλύτερο. Αλλά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε κρίση. Να έχει δηλαδή τα αρχικά στοιχεία στη διάθεσή του. Αν για παράδειγμα πείτε, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ότι θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο αλφαβητισμού. Θα πρέπει να πούμε ποιο είναι το επίπεδο αλφαβητισμού αυτή τη στιγμή. Και από τη στιγμή που ξέρουμε ποιο είναι το ισχύον και έχει γραφτεί αυτό στο έγγραφο της Κομισιόν, μπορούμε να κάνουμε και μια πρόταση, ένα στόχο σε σχέση με αυτό που ισχύει τώρα. Αλλά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να κρίνει να έχει δηλαδή τα στοιχεία, τα αρχικά, την κατάσταση δηλαδή πώς έχει τη στιγμή πριν από την απελευθέρωση των χρημάτων για να μπορούμε να κρίνουμε μετά αν υπάρχουν στοιχεία, με νούμερα αν είναι αυτό δυνατόν. Απτά. Γι' αυτό λοιπόν να δίνουμε αυτό το παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Η συγγήτρια μας θέλει κάτι να πει, να κλείσει. Όχι. Ωραία. Εφόσον δεν υπάρχει κανείς άλλος που να έχει το λόγο, να προτείνω να κλείσουμε το 4 της ημερήσιας διάταξης και να πάμε στην εξέταση του 5, που είναι μια παρουσίαση πρόοδου όσον αφορά την μεταρρύθμιση της υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης. Και ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν στην προηγούμενη συζήτηση και δίνω το λόγο την εισηγήτριά μας, κυρία Ίγκερ Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχω πολύ χρόνο ομιλία σήμερα, υπερβολικό, αλλά πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είχε αναβληθεί την προηγούμενη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Πρόκειται για μια ενημέρωση της ε, τελευταίας ε, διαδικασία ε, του Όλαφ. Μετά από πέντε τριμερείς διαλόγους που σαν ολόκληρη ημέρα, και ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Έχουμε περάσει στο 13α πλέον, στο άρθρο 13α. Άρα δεν μας μένει πολύ μέχρι το τέλος πλέον. Τα έχουμε όλα πλέον στη διάθεσή μας. Ε. Έχουμε τον αναφερειμένο κανονισμό πλέον. Και έχουμε βάλει τα στοιχεία με τους παχιούς χαρακτήρες αυτά που έχουμε συμφωνήσει και τέλος έχουμε αφήσει αυτά που λείπουν. Δεν έχουν μείνει πολλά με αχνούς χαρακτήρες, αλλά έχουμε το παράδειγμα 1 που λείπει. Επίσης, ε, από το παράδειγμα 1 μάλλον λείπουν σημαντικά κομμάτια. Να δώσω λίγο μια εντύπωση για το πώ έγιναν οι συζητήσει μέχρι τώρα. Τα βασικά προβλήματα δεν τα έχουμε με το Συμβούλιο, αλλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε με την Όλαφ, αλλά με τη Γενική Γραμματεία. Το θέμα λοιπόν το οποίο θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό είναι κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για μια ανεξάρτητη Όλαφ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, απόπειρες ε, να προσβληθεί από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ανεξαρτησία της Όλαφ. Αυτό θα το θέσω και στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Η Όλαφ τώρα δείχνει διάθεση συνεργασίας τη συζητήση, Αλλά αν είχαμε μόνο την Όλαφ για να συζητήσουμε, όπως σας είπα, θα είχαν τελειώσει προπολού οι διαπραγματεύσει. Τα δύο τρίτα των συζητήσεων γίνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη Γενική Γραμματεία. Για το παράδειγμα ένα τώρα, από αρχή μέχρι τέλου. Έχουμε ένα πρόβλημα ορισμού. Δεν μπορέσαμε ω τώρα να συμφωνήσουμε για το τι θα κάνουμε με τον όρο ατασταλίες. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις ε, αρμοδιότητες της υπηρεσίας στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει ε, οποιαδήποτε σαφήνεια ότι η Όλαφ είναι υπεύθυνη για τέτοιες ατασταλίες. Εμείς προσπαθ... μάλλον οι προσπάθειε μας να οριστούν αυτές οι αρμοδιότητες στον κανονισμό δεν έχουν στεφτεί ακόμα με ε, επιτυχία και σε αυτό το σημείο είναι πολύ αποφασιστική και η στάση του, του Συμβουλίου. Το Economic Operators Involved Indirectly, οικονομικοί φορεί που εμπλέκονται έμεσα. Το θέμα δηλαδή του ποιου μπορεί να ελέγχει, ποιο μπορεί να ελέγχει η υπηρεσία σε ό,τι αφορά επίσης ε, τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας για το Memorandum of Understanding. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει να μην είναι δεσμευτικά, ε, δεσμευτικές οι συμφωνίες. Ε, αν το γράψουμε αυτό, τι νόημα έχει να συνάψουμε οποιαδήποτε συμφωνία εφόσον δεν είναι δεσμευτική. Αυτό θα αναφερθεί σε τελογική σκέψη. Ανοιχτό είναι ακόμα το θέμα των δικαιωμάτων της Όλαφ για τα γραφεία των βουλευτών και κυρίως για τους βοηθούς. Αύριο το πρωί θα γίνει μια προπρασκευαστική συνάντηση και πολύ θα χαρώ αν στη συνάντηση αυτή καταφέρουμε να συζητήσουμε και με τους κοιόδης πώς θα ρυθμιστεί το θέμα αυτό. Έχουμε επίσης ένα θέμα προστασίας δεδομένων και σε ό,τι αφορά την ε, υπηρεσία τη σχετική της Ευρωπαϊκής Ένωση. Το θέμα είναι ποια είναι η πρόσβαση που πρέπει να έχει όλα στα προσωπικά αυτά δεδομένα. Ένα βασικό εκκρεμές ζήτημα για τα ε, δικαιώματα των συμμετεχόντων των, ε, στο εσωτερικό της Όλαφ. Ποια θα πρέπει να είναι. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει τίποτα γιατί έχει καταστεί σαφές ότι αν κάποιος κατά τη διάρκεια μιας έρευνας Όλαφ κάνει μια καταγγελία και θελήσει να διευκρινιστεί η κατάσταση στην Όλαφ, είναι ένα θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι θα το λύσουμε σύντομα. Βάση είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου. Υπάρχουν λίγα μόνο σημεία τα οποία δεν ε, καλύπτονται από τις τροπολογίες. Για παράδειγμα, τα θέματα της πρόσβασης στα γραφεία των βουλευτών. Τα θέματα αυτά, λοιπόν, αναφέρονται ξεχωριστά και θα, θα συζητηθούν αύριο, δύο εξ αυτών τουλάχιστον. Και το θέμα της ε, Επιτροπής Ελέγχου σε ό,τι αφορά την επικάλυψη θέσεων. Ε, παράλληλα διεξάγεται και η ομάδα υψηλού επίπεδου Υπάρχουν λοιπόν στο σημείο αυτό ε, θέματα που αλληλοεπικαλύπτονται, όπως για παράδειγμα τα θέματα της, ε, των θητιών που ε, παρουσιάζουν επικάλυψη. Δεν προβλέψαμε τέτοια διαδικασία στις τροπολογίες μας. Εργαζόμαστε με απόλυτα διαφανή τρόπο, δεν υπάρχουν μυστικά για τίποτε. Αλλά πολύ θα εκτιμούσα αν υπό την Πολωνική Προεδρία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τη Εγώ έχω μεγάλη θεσιμότητα, τους έχω δώσει και πάρα πολλές ημέρες που είμαι διαθέσιμη. Εκτός και αν δεν είναι πλέον τόσο αισιόδοξη η Πολωνική Προεδρία ότι θα τα καταφέρει αν έχει χάσει λίγο ε, την αισιοδοξία της. Ε, να παρακαλέσω λοιπόν την Πολωνική Προεδρία να ολοκληρώσουμε το, τη διατύπωση. Το Συμβούλιο έχει ορίσει συμβούλιο συνάντηση 6 Δεκεμβρίου. Θα πρέπει να το συζητήσουμε σίγουρα αυτό μετά τις 6 Δεκεμβρίου, γιατί είναι καταπήγον το θέμα αυτό. Να παρακαλέσω λοιπόν το Συμβούλιο να συνεχίσουμε τις εργασίες για να καταλήξουμε σε ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Θα προσπαθήσουμε τα εκκρεμή ζητήματα τα οποία είναι εσωτερικά δικά μας να τα διευκρινίσουμε σε ό,τι αφορά τη διατύπωση. Να παρακαλέσω λοιπόν τους συναδέλφου τους κοιότες να έρθουν στι 9. Είναι πραγματικά απαραίτητο. Πρέπει να λάβουμε κάποιες απαντήσεις, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτά ήθελα να πω. Merci. ευχαριστώ. Ο Καταρχήν, θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ τη συνάδελφο Γκρέσλερ για την ισχυρή θέση που καταλαμβάνει η του, του Συμβουλίου και της Κομισιόν και ευχαριστώ επίσης για την ε, διαφάνεια και μιλώ και εξ ονόματος του Σκιώδου της ομάδας μου του κ. Σκυλακάκη ποιος θεωρεί πραγματικά τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, όσον αφορά τον ορισμό των ε, οικονομικών συμφερόντων, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να βρούμε μία λύση για έναν ορισμό που να είναι πολύ ευρύ, κυρία Γκρέσλε. Το Δεκέμβριο ίσως θα έχουμε τις πρώτες ε, προτάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ε, μεταρρύθμιση της συνθήκης. Θα έχουμε μια αφορολογική ένωση, θα έχουμε μια οικονομική ένωση. Ποια θα είναι η αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε νέες ευθύνες για την Όλαφ. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις προτάσεις. Είχαμε μια συζήτηση τι θα κάνουμε με, το, ε, με τα διάφορα ταμεία και υπό το φως αυτών θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Δεύτερον, το θέμα της πρόσβασης στα γραφεία των βουλευτών. Υπήρχαν διάφορες υποθέσεις και η πιο χαρακτηριστική είναι του συναδέλφου Σάλμπα που είχε τύχει παρεμίων επιθέσεων από τα άλλα Σεβερίν κλπ. Και εκείνος ζήτησε να δράσει η Όλαφ σε αυτή την περίπτωση και μέσω εκείνου είχε πρόσβαση στο γραφείο του η Όλαφ και αυτό οδήγησε σε γλίγορη διευκρίνηση της υπόθεσης. Νομίζω ότι αυτός ο εκούσιος χαρακτήρας θα είναι κάτι που θα πρέπει να διατηρηθεί. Δηλαδή, αν επιθυμεί συνεργασία με την Όλαφο η θα πρέπει κάτι τέτοιο να είναι δυνατό. Υπάρχουν κάποιε αμφιλεγόμενε υποθέσει. Ξέρω ότι το Προεδρείο, ιδίω ο Γενικό Γραμματέα, έθεσε το θέμα στο θέμα αρχή. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή ευρωπαϊκή συγγελία, δεν, υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση, αλλά αυτή η ρήτρα δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία εμποδίων πραγματικά. Δεύτερον, η Εποπτική Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση περί τίνο πρόκειται και το θέμα των επικαλύψεων. Αν νομίζω ότι για τη σημεία αυτό θα πρέπει να έχουμε τη δομή κατά νου, όχι τη μικροδιαχείριση. Αν έχουμε δηλαδή τη σωστή δομή, δεν θα πρέπει να μπλεχθούμε με λεπτομέρειες. Εύχομαι όμως κάθε επιτυχία στη συνάδελφο Γκρέσλε και πολύ δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Γκρέσλε για την εργασία της εν την ε, μεταρρύθμιση αυτή. Είναι μια εργασία πολύ ουσιαστική και ορισμένα θέματα πραγματικά παρουσιάστηκαν σαν ε, προβληματικά, όπως ας πούμε αυτό με τα γραφεία των βουλευτών. Υπάρχει ένα θέμα αρχής ε, του Όλαφ. Πρόκειται για προστασία εκείνων των ατόμων φυσικών και νομικών ατόμων για τα οποία έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαδικασία αφενός και αφετέρου οι προθεσμίες είναι όσο πάει και πιο μακρές για τις διαδικασίες αυτές. Η διάρκεια των διαδικασιών, δικαστικών διαδικασιών και άλλων είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα γιατί εκεί μπορεί να καταστραφεί μια υγιής δημοκρατία. γιατί σε αυτό το κενό στο οποίο εργαζόμαστε και στο οποίο τοποθετείται και η όλα και όπου υπάρχουν τόσες πολλές αμφιβολίες για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές να ε, βρουν μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση. Δηλαδή, εσωτερικό θέμα μόνο για το κοινοβούλιο δεν νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί οι εκπρόσωποι του ΟΛΑΦ θέλουν να προασπίσουν τη δική τους ε, υπηρεσία, το δικό τους ε, όργανο. Εκεί είναι η μόνη υπηρεσία που μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητες προφορές και δεν θέλουμε να εμπλακεί σε πολύπλοκες καταστάσεις η Όλαφ. Την περαιτέρω έκθεση ανεβλήθηκε και θα ήθελα να παρακαλέσω την εισηγήτρια τώρα να μιλήσουμε ανοιχτά. Να πει η εισηγήτρια, δημόσια. Ανησυχούμε. Βέβαια θα πρέπει να διατηρήσει την ανεξαρτησία της η Όλαφ, αλλά οι αλλαγές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή που πραγματοποιούνται για την Όλαφ αυτή τη στιγμή δεν σημαίνουν ότι θα πρέπει να έχουμε ε, αυτή την υπηρεσία που θέλαμε που θα υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία της Όλαφ όχι, γιατί εδώ δημιουργούνται και άλλες δυνατότητες. Λες και πρόκειται για δικηγόρους. Ενώ πρόκειται για τον κεντρικό πυλώνα των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. Και γι' αυτό δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την εισηγήτρια. Λέγοντας ότι εγγυήσεις των διαδικασιών αυτών και το γεγονός ότι θα πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι ότι παίζει το συγκεκριμένο της ρόλο η Όλαφ εκ παραλίλου προς την Κομισιόν που ασχολείται με στατιστικά κλπ ότι υπάρχει ε, μια συγκεκριμένη και σημαντική αξία για την Όλαφ. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι κάπως είμαστε το Συμβούλιο της, ε, της ε, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να είναι εξάρτητη η υπηρεσία αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το έγγραφο για την μεταρρυθμίση της Όλαφ είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας μετά από ότι θέση σε τη της Συνθήκης Λισαβόνας. Ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα. Να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια, την Ίγκεμπορ που ανέχτηκε όλες μου τις απουσίες της διαπραγματεύσεις για υποκειμενικούς και αντικειμενικούς λόγους, αλλά όπως σωστά αναφέρθηκε, το βασικό θέμα είναι πώς θα διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της Όλαφ. Προκειμένου να λαμβάνουμε εύκολα πληροφορίες και να δίνουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις που μας τίθενται για την καλή χρήση των πόρων. Στο προηγούμενο θέμα το συζητήσαμε εκτεταμένα και οι βασικές λειτουργίες της Όλαφ είναι σαφείς και οι βασικές αρχές. Όλοι συμφωνούμε ότι τα όσα έχουμε πετύχει είναι θετικά. Και νομίζω ότι και η ίδια η Όλαφ το αντιλαμβάνεται αυτό, το αντιλαμβάνεται επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Όλαφ θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να έχει δικαίωμα σε πρόσβαση και συλλογή δεδομένων, στοιχείων θα πρέπει να έχει πολιτικούς αξιωματούχους οι οποίοι θα μπορούν να αποφασίζουν για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνεται και η ανεξαρτησία αφετέρου θα πρέπει να περιορίζεται με τέτοιο τρόπο προκειμένου τα θεσμικά, το θεσμικό όργανο και τα θεσμικά όργανα να εκπληρώνουν τις ε, αρμοδιότητες του σε ό,τι αφορά την έρευνα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στα 11 άρθρα και στα θέματα των ε, διαδικαστικών εγγύησεων. Νομίζω ότι η πρόταση γενικά είναι καλή. Θα πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τις δικαστικές αγωγές και θα πρέπει να φροντίσουμε στη διαδικασία αυτή, όπως είπε και η ίδια η να ε, καταλήξουμε σε τελική συμφωνία επί του τελικού κειμένου υπό την Πολωνική Προεδρία και η Όλαφ στο μέλλον θα έχει μια καλύτερη, ένα καλύτερο ορισμό, μια καλύτερη δομή εντός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πεδίο αυτό αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών και των κρατών μελών, την Eurojust, την Europol, τα Υπουργεία, τα σχετικά με την ασφάλεια στα κράτη-μέλη, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι και καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Η Κομισιόν προσέλαβε δύο λόγια. Όχι. Δεν θέλετε να, να την ώρα. Ε, βέβαια, άμα θέλετε να σας πούμε δύο λόγια. Είναι απόλυτα ευτυχή η Κομισιό να συνεργάζεται με την κυρία Γκρέσλε και το Συμβούλιο για να βελτιωθεί ο κατεβός 1703. Ε, η Κομισιόν ήδη είχε υποβάλει αυτή την πρόταση. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με πνεύμα συνεργασίας ε, στεναχωρέθηκα να ακούσω την κυρία ε, Γκρέφλε που είπε ότι το εμπόδιο στη διαπραγματεύση είναι η Κομισιόν. Εγώ δεν έχω την ίδια εντύπωση. Νομίζω ότι όλε οι υπηρεσίε προσπαθούν να πετύχουν το ίδιο στόχο, δηλαδή να υπάρχει με όλα ανεξάρτητη, αποτελεσματική και με διαδικασίες σαφείς. Και γι' αυτό θεωρούμε, ελπίζουμε μάλιστα, ότι το, ο κανονισμός θα έχει τα πιο αυστηρά ε, κριτήρια, ιδίως όσον αφορά τις εγγύσεις των ε, αγωγών, για να μην χρειαστεί να υπάρχει μια άλλη νομοθεσία που ορίζει κάποιες λεπτομέρειες των διαδικασιών αυτών για τις άγωγες. Ε, Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι μέσα στην, στον ίδιο κανονισμό. Αλλιώ θα υπάρχουν μόνο διακονισμοί των λεπτομέρειων. Λυπάται πολύ η Κομισιόν που δεν τα βλέπει τα πράγματα έτσι και η κυρία Γκρέσλε αλλά που δεν είδε έχει την πρόθεση η Κομισιόν να μειώσει την εξαρτησία τη όλα αυτούν αντίον. Ενδιαφέρεται όμω η Κομισιόν ε, για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων όλων των ατόμων, όλων των ε, θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών ενδιαφερόμαστε για την προστασία των βουλευτών και των βοηθών τους, αλλά θα πρέπει από την άλλη μεριά να μην ξεχνάμε ότι η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για το σύνολο της Ευρωπαϊκή για την προστασία των δεδομένων όλων των εμπλεκομένων. Αναζητούμε λοιπόν λύσεις, δεν ξέρω αν θα τις βρούμε στις επόμενες μέρες, αλλά θα συνεργαστούμε ε, με χαρά και πολύ ανοιχτά με την κυρία Γκρέσλε και με το Συμβούλιο. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την δήλωση αυτή προθέσεων. Η εισηγήτριά μας θέλει να πει κάτι. Η εκπρόσωπος της Όλαφ έχει να πει κάτι. Μάλιστα. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα πράγματι να τονίσω αυτά που ελέγχθησαν για πραγματική ανεξαρτησία της Όλαφ μέσα στις πλαίσια διαδικασιών και αγών είναι πάρα πολύ σημαντική. Και μια που έχει διαθεσμική αρμοδιότητα η Όλαφ είναι αυτό πρωτή σημασία. Θα ήθελα να τονίσω λιγάκι αυτό που ελέγχθη ότι ξεκίνησε δηλαδή ο τριμελής διάλογος σε πολύ επικοινωνικό κλίμα, δεν νομοθέτης η Όλαφ. Εμείς συμμετέχουμε και προσπαθούμε να συμβάλλουμε θετικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχει διάσπευση από πολλές περιφέρειες για την επίτευξη λύσης και ελπίζω ότι αυτός ο δυναμισμός που ξεκίνησε χάρη στη θαυμάσια έκθεση του Κοινοβουλίου και στον δυναμισμό της σημερινής Προεδρίας θα συνεχίσει. Συμμερίζομαι λίγο τις ανησυχίες της κυρίας Γκρέσλε ότι δεν έχουμε απτά αποτελέσματα από την πολιτική πρόεδρια. Υπάρχει ο κίνδυνος παράτασης των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το των δυνατόν. Υπάρχει ένας ε, de facto μεταξύ αυτών Τη εξέτασης και αυτών που γίνονται εσωτερικά στην Όλαφ, που γίνεται μια αναδιάρθρωση της εργασίας. Ελπίζουμε λοιπόν οι διαπραγματεύσεις να μπορούν να στεφθούν από επιτυχία το γλυγορότερο δυνατόν και έχουμε, να έχουμε έτσι μια νομική ασφάλεια. Αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνει και τις εγγυήσεις για τις Δικασίε που ακολουθούν και για τις αγωγέ μέσα στα πλαίσια των ερευνών τη Όλαφ. Και θα πρέπει έτσι από κοινού να προσπίσουμε την αρχή των οικονομικών συμφερόντων και θα πρέπει να δώσουμε ένα ορισμό τον ευρύ. Ιδίως ε, λόγω των προσφάτων ε, θεσμικών εξελίξεων. Νομίζω λοιπόν ότι τα σημεία που μας χωρίζουν δεν είναι πόσο σημαντικά, όσο δυσκολίε μπορούμε να ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ κύριε Κό, λέει ο πρόεδρο. Η συγκήτρια θέλει να πει δύο λόγια για να ολοκληρώσει. Μια και καθόμαστε εδώ και τα λέμε ωραία, να πω κι εγώ κάποια σχόλια. Θα ήθελα να πω ότι δεν ήθελα να τρέξω το δόντια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασφαλώ, γιατί παντού θέλω να έχω φίλου. Αλλά θα ήθελα να πω ότι κάποια σημεία με έκανα να σκεφτώ ιδιαίτερα και να αμφισβητώ διάφορα πράγματα. Καταρχάς, ε, ενώ διαπραγματευόμαστε από κοινού και συζητάμε τη νέα δομή τη Όλαφ, την ιστορική δομή τη Όλαφ, ο Γενικός Γραμματέας ε, ε, ε, υποστηρίζει ένα οργανόγραμμα για την Όλαφ που δεν ταιριάζει καθόλου με την έκθεσή μας. Το θέμα λοιπόν που συχνά έχω θίξει για το πόσο σοβαρά λαμβάνεται η συναπόφαση. Κατανοώ ιδιαίτερα το ότι έχει ανώτερη αρμοδιότητα στα θέματα διοργάνωσης, οργανωτικά. Αλλά σε ό,τι αφορά ιστορικές διαδικασίες θα πρέπει να ξέρουμε το πώς, ποια είναι τα δικαιώματα του καθενός, γιατί αυτό επηρεάζει άμεσα την έκθεση και θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Και το θέμα δεν είμαι εγώ για να κάνουμε μια συζήτηση δυο Το θέμα είναι πώς θα βρούμε μια δομή που θα αποτυπώνει αυτά που θέλουμε. Αυτά αφενός. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Το δεύτερο θέμα για την ανεξαρτησία της Όλαφ. Μου λέτε ότι ο Γενικός ε, ε, Γραμματέας θέλει να είναι απίστευτα αυτά τα καινούργια κινητά και το δικό μου κινητό. με το συμπαθώ καθόλου. Για το IPN, για την ε, πρόσληψη, των διορισμό προσωπικού. Αν ε, αυτό πάυσει θα είναι κάτι που θα ανησυχήσει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την Όλαφ. Η γνωμοδότηση της Υποπτικής Επιτροπής για την διαδικασία αυτή. Ο Γενικός Γραμματέας ε, σε ό,τι αφορά τα non-cases, τις υποθέσεις που δεν ε, λαμβάνουν συνέχεια, όπου περιλαμβάνονται όμως όλα τα ονόματα αυτές οι περιπτώσεις ή αυτές οι υποθέσεις διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κυκλοφορούν λοιπόν αυτά τα ονόματα ανοιχτά. Θα ήθελα έκθεση ε, του Οργανισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Επίσης, ε, τα θέματα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Το θέμα, για παράδειγμα, του τι σημαίνει για την Όλαφ η μεταρρύθμιση του κανονισμού του καταστατικού για το προσωπικό, για τους υπαλλήλου. Δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα, για παράδειγμα, όσο δεν υπάρχει απόφαση. Αυτό το προβλέπει ο κανονισμός σε ό,τι αφορά τα πτραχικά μέτρα ε, πριν από την λήψη δικαστικής απόφασης. Γι' αυτό θα χρειαζόταν μια μικρή αλλαγή στο κανονισμό για να υπάρχει τέτοια δυνατότητα ίδιας ερέπνας. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με βαθιά προβλήματα. Ένα άλλο βαθύ πρόβλημα είναι η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε με το Συμβούλιο για το πόσο σημαντικό, σημαντικά ε, είναι τα θέματα καταπολέμησης απάτης στο Συμβούλιο. Το αυτό που είπε η συνάδελφος Αγέλα Σέντερ για το Procedural Code, τον κώδικα διαδικασίας. Να σας πενθυμίσω ότι το 2008 έγινε σχετική τροπολογία για το Procedural Code να συμπεριληφθεί στη συναπόφαση. Πολλές φορές το έχω δείξει το θέμα αυτό και φυσικά φαντάζεσαι ότι δεν με αντιμετωπίζουν με στοργή και αγάπη. Όταν καλούμαστε να συζητήσουμε τέτοια θέματα, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε εμείς μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα του κώδικα και θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Αυτό που είπε ο κ. Χατζημαρκάκης για την ε, χρηματοοικονομική ένωση, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά θα πρέπει να δούμε Μήπως πρέπει να αλλάξει ο ορισμός των οικονομικών συμφερόντων. Η Χρηματοπιστωτική Ένωση φυσικά ε, κατεστεί ακόμα πιο έντονη την ανάγκη αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση την οποία και με μεγάλη ενδελέχεια θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτά που είπε η κυρία Σέντερ για το θέμα της ανεξαρτησίας της Εποπτικής Επιτροχής. Μάλιστα, αλλά πρέπει να πω ότι πάντα πίστευα ότι όλα αυτά θα πρέπει να διοργανώνονται με ήρεμο τρόπο σε μια τέτοια υπηρεσία. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα αυτό δεν είναι εφικτό. το να προβλεφθούν τα συστήματα στον κανονισμό, συστήματα ε, ανεξαρτησίας προσωπικού και το καθεξής. Δεν έχουμε τροπολογίες στο σημείο αυτό. Θα πρέπει να τις ε, καταθέσουμε εκ των υστέρων. Θα βρω σε μια τέτοια διατύπωση. Θα τη συζητήσουμε αύριο το πρωί. Το έχω θίξει το θέμα αυτό και στο Στρασβούργο άλλωστε. Κατανοώ τα προβλήματα λοιπόν που υπάρχουν. Είμαι αισιόδοξη. Έχουμε τόσες πολλές συζητήσεις άλλωστε και είναι καλό το κλίμα των διαπραγματεύσεων. Το τονίζω αυτό. Άρα ναι, πραγματικά είμαστε όλοι φίλοι. Σας το ορκίζομαι. Και όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα, αν κάποιος ε, έχει διαφορετική άποψη από κάποιον άλλο για το ποιο είναι το καλό αποτέλεσμα, αυτό είναι θεμητό. Να ευχαριστήσω την γραμματεία που κάνει εξαιρετικό έργο και την κυρία Φαντζέλο, την δική μου ε, βοηθό θα ήθελα να ευχαριστήσω και κάποιους υπαλλήλους της ομάδας και κάποιους ε, γενναίους βοηθούς. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο αυτό, δεν μπορώ όμως και εγώ να το αλλάξω. Να έχετε υπομονή όμως και θα ολοκληρωθεί. Merci. La commission, euh, Madame Ευχαριστώ. Η Κομισιόν ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Μισό δευτερόλεπτο. Έχει σχέση με ένα ίσονο σημασία θέμα, το οποίο έθιξε η κυρία Γκρέσλε, το οποίο ωστόσο είναι σημαντικό και αφορά την αποστολή των τελικών εκθέσεων που έχουν κλείσει και που δεν χρειάζεται να γίνεται, να δοθεί συνέχεια και που η κυρία Γκρέσλα ανησυχεί πως υπάρχει πρόβλημα προστασίας των ε, όσων ε, ενημερώνουν. Εμείς τακτικά ζητάμε από την Όλαφ και από τον ΤΠΕΣ, το έχει ζητήσει, τα ονόματα να μην αναφέρονται στις τελικές εκθέσεις, είτε αυτές είναι για να δοθεί συνέχεια είτε όχι. Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρονται τα στοιχεία αυτά στις εκθέσεις και έχουμε θυμίσει στην Όλαφ ότι μόνο κατ' εξαίρεση το άρθρο 9.4 του ισχύοντος κανονισμού προβλέπει ότι οι εκθέσεις και τα σχετικά έγγραφα θα σταλούν στο θεσμό, σώμα ή υπηρεσία το ενδιαφερόμενο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η Κομισιόν που το λαμβάνει. Κάθε θεσμικό όργανο, body, σώμα ή υπηρεσία θα πρέπει να λαμβάνει τελική έκθεση. Και γιατί. Διότι Ακόμα και αυτές οι εκθέσεις όπου δεν δίνεται συνέχεια μπορεί να οδηγήσουν στη λήψη διοικητικών μέτρων, στη βελτίωση της διαχείρισης. Δεν σημαίνει ότι μια έκθεση που κλείνει χωρίς να δοθεί συνέχεια δεν έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την βελτίωση της ε, οικονομικής διοίκησης. Θα ήταν λοιπόν ε, κακό και δεν προβλέπεται να πετάγεται οποιαδήποτε έκθεση που έχει κλείσει χωρίς να της δοθεί συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό, προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν προβλέπεται τροποποίηση. Γιατί αντίθετα Όλα τα θεσμικά όργανα, οι υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται. Και δεν είναι θέμα διάδοσης των πληροφοριών, γιατί μια τελική έκθεση που θα κλείσει χωρίς να δοθεί συνέχεια θα παραμείνει ε, απόρριτη. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την καλύτερη περάσπιση των οικονομικών συμφερόντων. Ευχαριστώ. Η συγκέντριά μας θέλει να κλείσει. Λυπούμε, ναι, είμαι αναγκασμένη να επανέλθω. Αναφέρομαι στη γνωμοδότηση υπ. 5 που συστήνω σε όλα τα μέλη να την διαβάσουν. Γιατί εδώ η Επιτροπή Επιτήρησης αναφέρεται, αν δεν κάνω 38 υποθέσεις που έχει εξετάσει. Υπάρχουν λοιπόν οι φάκελοι, γιατί έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι υποθέσεις, αλλά θα είχαν μπροστά τους το περιεχόμενο και στη γνωμοδότηση είναι ότι υπάρχουν αναλυτικές αναλυτικά στοιχεία που επιτρέπουν να μπορέσει κανένας να αναπλάσει το ποιος ήταν ο υπεύθυνο και τι έγινε. Το θέμα ότι το είχαν τα, τα, τα παίρνει τα στοιχεία αυτά η Κομισιόν και όλε τι άλλε υπηρεσίε είναι ότι υπάρχει ένα είδη clearing house μεταξύ Όλαφ και επιτροπή. και έτσι παίρνει τι πληροφορίε αυτέ η Κομισιόν και μετά δίνονται και στι άλλε υπηρεσίε. Γιατί άμα ξέρει κανένα ποιο διαχειρίζεται τα εν λόγω ταμεία, μπορεί κανένα αμέσω να καταλάβει ότι αυτό αφορά την Κομισιόν άμεσα. Ελπίζω ότι έχουμε ένα κοινό συμφέρον που σημαίνει ότι παίρνουμε κάποιες ενδείξεις και ακολουθούμε. Ότι υπάρχει κάποιο, κάποιο πρόβλημα και νομίζω ότι αυτό είναι μια επικίνδυνη υπόθεση στην, στην, στην Ένωση αυτό με αυτούς που προειδοποιούν τους whistleblowing είναι λοιπόν σημαντικό το θέμα αυτό. Θα πρέπει να το εξετάσουμε γιατί αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Η Επιτροπή ε, Επιτηρήσεις λέει ότι η αρχή της ανάγκης του να γνωρίζει κανένας περί τίνος πρόκειται καταπατάται συνεχώς. Συστηματική πρόθεση δηλαδή των στοιχείων είναι σημαντική. Αύριο το πρωί έχουμε ε, πάλι συνάντηση. Εγώ ε, κάθε Κυριακή βράδυ είμαι στις Βρυξέλλες. Ε, αφού σας έχω εσάς, τι άλλους φίλους χρειάζομαι. <laughs> Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γλίγορα βέβαια με τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ για την ολοκλήρωση αυτή. Κανένα άλλο δεν ζητάει το λόγο. Προτείνω να κλείσουμε λοιπόν το σημείο 5 τη διάθεση, Το 6 αναβλήθηκε απουσία του ε, εισηγητή του κυρίου Μπαλτεστά. Αν κανένα άλλο δεν θέλει το λόγο, διακόπτει η συνεδρίαση μέχρι το απόγευμα. Τρει στην ίδια